Okay. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθατε εδώ σήμερα το απόγευμα. Φαντάζομαι και άλλοι ευρωβουλευτές ε, θα φτάσουν, ίσως λίγο καθυστερημένα, αλλά ας αρχίσουμε. Καλωσορίζω την κυρία Ναμαρ Χάριξον, που είναι Υπουργό Δικαιοσύνη τη Φιλανδία, για να μα παρουσιάσει το πρόγραμμα τη Φιλανδική Προεδρία για τα θέματα που μας αφορούν. Να σας δώσω το λόγο για 15 λεπτά για την παρουσίασή σας και μετά να ακούσουμε ερωτήσει από τους ευρωβουλευτές. Συμφωνείτε? Ωραία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Λούση Νέτσιγκα, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα ενώπιον σας για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκλογές της άνοιξη, οι ευρωπαϊκές εκλογές, ήταν ε, σαφώς μια ψήφος εμπιστοσύνης υπέρ της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Η αυξημένη συμμετοχή του κόσμου στις εκλογές αυτές έδειξε ότι οι άνθρωποι νοιάζονται, πιστεύουν στην Ευρώπη και θέλουν η Ευρώπη να έχει έναν ισχυρό ρόλο για να αντιμετωπιστούν οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Έτσι λοιπόν, με υψηλές προσδοκίες και με όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, σημαίνει ότι συγχρόνως έχουμε και μεγαλύτερες ευθύνε. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες αυτές, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω απ' όλα μια κοινότητα αξιών. Και ακριβώς αυτή η κοινή μας ε, βάση αξιών είναι που μας καθιστά ισχυρούς. Το φιλόδοξο σλόγγαν της Φιλανδικής Προεδρίας είναι «Βιώσιμη Ευρώπη, βιώσιμο μέλλον». Έτσι λοιπόν μαζί πρέπει να εργαστούμε για να ενισχύσουμε τις κοινέ μας αξίες και το κράτος δικαίου. Μαζί πρέπει να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο ανταγωνιστική με τη συμμετοχή όλων Πρέπει να ενισχύσουμε την θέση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ως ε, παγκόσμιο ηγέτη σε θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική δράση και να διασφαλίσουμε βέβαια και την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών. Όσον αφορά την πρώτη προτεραιότητα, δηλαδή να διασφαλίσουμε και να ενισχύσουμε τις κοινέ μας αξίες και το κράτος δικαίου. Αυτό αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο για όλες τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί επηρεάζει κάθε πτυχή, τόσο τα θεμελιώδη δικαιώματα, όσο και την ε, καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Παραβιάσεις στο κράτος δικαίου υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων όσον αφορά τα δικαιώματά τους. Διστάζουν να πιστέψουν τότε ότι προστατεύονται τα δικαιώματά τους και να εμπιστευτούν το ευρωπαϊκό σύστημα. Το κράτος δικαίου λοιπόν, πολύ ορθά, αποτελεί με από τις κύριες προτεραιότητες των νέων ευρωπαϊκών στόχων στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και της νέας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Σούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να ενισχύσουμε τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ του κράτους δικαίου. Η Φιλανδία λοιπόν χαίρεται και καλωσορίζει την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και για τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού ετήσιας ε, αναφοράς. Έχουμε δεσμευτεί να προχωρήσουμε με συγκεκριμένους ε, στόχους όπως αναφέρονται και στην ανακοίνωση του Συμβουλίου. Θέλουμε ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια. Αυτό είναι στην καρδιά του κράτους δικαίου εξάλλου. Και κάθε δικαστήριο το οποίο ε, δικάζει βάση του κοινοτικού δικαίου είναι και ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό όλες οι χώρες μέλη να φροντίσουν να διασφαλίσουν ότι το κράτος δικαίου θα προστατεύεται και θα τηρείται στις χώρες μας. Τον Ιούλιο ε, συγκάλεσα μία άτυπη συνάντηση των Υπουργών Δικαιοσύνης προκειμένου να συζητήσουμε την αρχή αυτή του κράτους δικαίου με στόχο να ενισχύσουμε τα μέσα που διαθέτουμε, την εργαλειοθήκη που διαθέτουμε και στον τομέα της δικαιοσύνης. Μέσα λοιπόν όπως είναι κοινή κατάρτιση των επαγγελματιών νομικών, στήριξη της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να προωθείται εκεί η νοτροπία του δικαίου και η ενίσχυση του βαθμολογίου όσον αφορά την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη είναι κάποια παραδείγματα. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να προωθήσουμε το κράτος δικαίου και μέσω της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μέλη της Επιτροπής Δικαιοσύνης. Τώρα τον Οκτώβριο θα έχουμε 20 χρόνια από τότε που συνεδρίασε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην φιλαδική πόλη του Τέμπερε προκειμένου να ξεκινήσει η ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Ο στόχο που τέθηκε στο Τάμπερε τότε ήταν ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να προσεγγίζουν τα δικαστήρια και τι δικαστικέ αρχέ σε οποιαδήποτε χώρα μέλη, σαν να βρίσκονται στη δικιά του. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποφασίσει από κοινού ε, για διάφορες ρυθμίσεις οι οποίες όντως προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών και ενισχύουν την δικιά τους νομική προστασία όταν κυκλοφορούν στην Ευρώπη, όταν ζουν κάπου αλλού στην Ευρώπη, εργάζονται ή φτιάχνουν την οικογένειά τους αλλού στην Ευρώπη. Πολλά έχουμε πετύχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν προβλέπει διατάξεις όσον αφορά την δικαιοδοσία των δικαστηρίων και την αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων. Έχουμε κάνει πολλά για να φτάσουμε στην αναρμόνιση κανόνων σχετικά με το δίκαιο και έχουμε βελτιώσει επίσης και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες. Και έχουμε αναπτύξει και σημαντικά εργαλεία και για την διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εθνικών δικαστικών αρχών σε θέματα αστικού δικαίου. Τώρα, στο μέλλον. Η τεχνολογική πρόοδος, η ψηφιοποίηση είναι πράγματα που επίσης θα παίξουν ρόλο κλειδί στον τομέα της δικαιοσύνης, γιατί μπορούν να συνεισφέρουν στο να επιταχύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Κατά τη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας, λοιπόν, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να μεταρρυθμίσουμε το θέμα των αποδεικτικών στοιχείων και την ρύθμιση που αφορά τα έγγραφα προκειμένου το Συμβούλιο να εγκρίνει μια γενική προσέγγιση κατά τη διάρκεια ακόμα της δικής μας Προεδρίας. Η νομική βεβαιότητα είναι κάτι πολύ βασικό και για τους πολίτες αλλά και για το διεθνές εμπόριο. Και όχι μόνο μέσα στην ενία αγορά, αλλά και εκτός συνόρων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μία τάξη για το εμπόριο, η οποία βασίζεται σε διεθνείς κανόνες, έχει περάσει από πολύ κριτική τα τελευταία χρόνια. Αλλά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την πολυμερή προσέγγιση. Η σύμβαση της ε, Χάγης που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι αποτελεί ένα καλό παράδειγμα πραγμάτων που έχουμε πετύχει στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας στη δικαιοσύνη. Η δεύτερη προτεραιότητα τώρα της Φιλανδικής Προεδρίας είναι μια ανταγωνιστική Ευρώπη με τη συμμετοχή όλων. Η ενή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Και το πιο σημαντικό μέσο για να βελτιώσουμε την ε, ανάπτυξη και την ευημερία είναι να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς. Και μπορούμε να έχουμε μια ισχυρή οικονομική βάση εμβαθύνοντας περισσότερο και ενισχύοντας τις τέσσερις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς. Πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της ψηφιακής επανάστασης, η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα και ε, πλατφόρμες οικονομίας είναι στοιχεία κλειδί για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης, της ευημερίας και της απασχόλησης. Η Νομική Επιτροπή έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο έργο αυτό που έχει να κάνει με νομικά ζητήματα όπως αυτά σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. Η Επιτροπή αυτή επίσης παίζει σημαντικό ρόλο προκειμένου να βαθύνουμε περισσότερο ακόμα στην ενία αγορά και να την καταστήσουμε περισσότερο αποτελεσματική. Το εταιρικό δίκαιο, η νομοθεσία που έχει να κάνει με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για την σημαντική της συνεργασία και για το ότι μας έχει βοηθήσει να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για πολλά ε, σημαντικά νομοθετικά ζητήματα και νομοθετικούς ε, φακέλους. Μαζί λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε ένα δίκαιο και προβλέψιμο πλαίσιο μέσα στο οποίο δρούν οι επιχειρήσεις. Η στενή συνεργασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει να αναλαμβάνουμε δράση για να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως είναι η φοροδιαφυγή και να μειώσουμε ε, καταστροφικές ε, συνέπειες από τον ανταγωνισμό στη φορολογία. Μαζί πρέπει να βρούμε τρόπους να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Χρειαζόμαστε μια δίκαια εσωτερική αγορά, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Θα συνεχίσουμε λοιπόν εργαζόμαστε για να ολοκληρωθεί ε, η νέα συμφωνία για τους καταναλωτές, το New Deal. Στόχος μας είναι το Συμβούλιο να καταλήξει σε μια γενική προσέγγιση όσον αφορά ε, οδηγία για δράσεις. Πρέπει να υπάρχει ένα ισορροπημένο σύστημα το οποίο στην πράξη να μπορεί να λειτουργήσει. Τώρα θέλω να επιστρέψω στην αρχή της ε, ομιλίας μου και να πω λίγα λόγια ακόμα όσον αφορά τις προσδοκίες των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών μας για να πετύχουμε διαφάνεια, ε, χρηστή δίκηση και καλύτερη νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Χρειάζεται σαφής επικοινωνία, περισσότερη διαφάνεια στις διαδικασίες ε, λήψης αποφάσεων, κάτι το οποίο μπορεί να φέρει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους πολίτες, να ενισχύσει τη δημοκρατία και να καταπολεμήσει την παραπληροφόρηση. Η χρηστή δίκηση και η διαφάνεια επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Παρόλο που η διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενισχυθεί πολύ όλα αυτά τα χρόνια, παραμένει αρκετή δουλειά να κάνουμε ακόμα. Χρειαζόμαστε ρύθμιση υψηλού επίπεδου και ενημερωμένη γιατί είναι κάτι το οποίο επηρεάζει απευθεία την ανταγωνιστικότητα. Μια ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία λειτουργεί ικανοποιητικά μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων. Συνεπώ, σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά για το έργο σα και για την ευκαιρία που μου δώσατε σήμερα να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα της Φιλανδικής Προεδρίας. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία μαζί σας κατά τη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας, αλλά και μετά από αυτήν. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed, um, Anna Maya. It's... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε και πρέπει να σας πω ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ αυτά που είπατε ε, σχετικά με τις φιλοδοξίες της ε, Φινλανδικής Προεδρίας. Πρώτη ερώτηση, κύριος, ε, κυρία, κυρία λέει η πρόεδρος, κυρία Βάλτσμαν, συγγνώμη που σας είπα κύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ε, παρουσιάσατε τις, ε, τα βασικά στοιχεία της Φινλανδικής Προεδρίας. Πράγματι, πολύ φιλόδοξη η στόχη σας. Χτες μπόρεσα να ανακοινώσω στον συνάδελφό σας, τον κύριο Ράκα, ότι όσον αφορά το ε, πρόγραμμα της ε, Φινλανδικής Προεδρίας. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει και το θέμα της ε, τεχνητής νοημοσύνης. Και εσείς αναφέρετε και την ψηφιοποίηση, την πλατφόρμα δεδομένων. Από πλευράς της δικής μας Επιτροπής θεωρώ ότι Πράγματι, αυτά είναι όλα πρόκληση. Καλούμεθα να καθορίσουμε ένα πλαίσιο. Και με όλα αυτά φτάνω στην ερώτησή μου, γιατί πρόκειται για ένα θέμα ε, όχι μόνο ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αλλά και προσανατολισμένο στο μέλλον. Και γι' αυτό το λόγο και εσείς ε, χρησιμοποιείτε αυτό τον όρο, το μέλλον που μπορεί να υπάρχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία, αλλά και για τους ε, πολίτες. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν υπάρχει το απαραίτητο πλαίσιο και ως εκ τούτου λείπει και αυτή η επένδυση και αυτή την αγορά δεν πρέπει να την αφήσουμε στα χέρια των Αμερικανών και της ε, Κίνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την τεχνολογία που διαθέτει θα πρέπει να συστήσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Βεβαίως για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και αυτό σημαίνει όχι να απαντάμε μόνο σε δεοντολογικά, σε θέματα δεοντολογικής φύσεως, αλλά και νομικής φύσεως, ε, σχετικά με τη χρήση, παραδείγματος χάρη των δεδομένων και τις ευθύνες που συνοδεύουν τα δεδομένα. Ερωτώ λοιπόν πολύ συγκεκριμένα. Κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας σας ε, έχετε συγκεκριμένα μέτρα κατά νου για το πώς θα προάγετε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εντάσσετε η τεχνητή νοημοσύνη που θα συνδυάζεται και με αυτά τα τρία προαναφερθέντα στοιχεία. Σας ε, εύχομαι επιτυχία, καλή επιτυχία από κοινού με τους συναδέλφους σας για να μπορέσετε να επιτύχετε τους στόχους σας. Θα, κάνουμε, θα δεχτούμε κάποιες ερωτήσεις και μετά ε, θα επανέλθουμε στην κυρία Υπουργό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας ε, και πριν και εγώ υποβάλω την ερώτησή μου, σας εύχομαι ειλικρινά κάθε επιτυχία στο φιλόδοξο πρόγραμμά σας. Και θα ήθελα πάρα πολύ ή χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα ε, αυτά που είπατε για το κράτος δικαίου και μια δίκαιη κοινή αγορά. Αυτό βέβαια ε, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Ένα εξ αυτών είναι η διαφάνεια, η ποικιλομορφία, η εκπροσώπηση σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Εμένα με ενδιαφέρουν οι εταιρείε και η οδηγία περί των δύο φύλων που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Συμβούλιο. Νομίζω είμαι σίγουρη μάλλον, ότι όλοι μας εδώ επιθυμούμε καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις εταιρείε, όχι μόνο στην πολιτική. Ε, το να υπάρχει μια ποικιλομορφία ε, στα διοικητικά συμβούλια, αυτό ε, συμβάλλει στο να υπάρχουν καλύτερες και πιο επικερδείς αποφάσεις. Ε, θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή η οδηγία έχει κολλήσει στο Συμβούλιο και θέλω να ρωτήσω τι θα κάνει η Φινλανδική Προεδρία για να προχωρήσει αυτός ο φάκελος, αυτό το θέμα. Tack så mycket för väldigt goda frågor. Thank you very much for this question. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας και θα απαντήσω στα σουηδικά. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ καλές οι ερωτήσεις που ετέθησαν και θα ήθελα να ξεκινήσω με την ερώτηση της ε, κυρίας Βάλτσμαν, η οποία ερώτησε για την τεχνητή νοημοσύνη. Ε, αυτό είναι ένα ιδιαίτερα επίκαιρο ερώτημα και νομίζω ότι υπάρχουν ε, τεχνολογίες οι οποίες έχουν ε, σχέση με την χρήση της ε, τεχνητής ε, νοημοσύνης. Αυτό έχει αυξηθεί κατά πολύ και στον νομικό τομέα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξελιχθεί περαιτέρω και θα χρησιμοποιείται συνειδητά λαμβάνοντας υπόψη το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ως εκ τούτου, αυτό που ενδιαφέρει είναι και να υπάρχει εμπιστοσύνη ε, στην ε, τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ερώτημα. Υπάρχουν πολλά ε, νομικής φύσεως θέματα που συμβαδίζουν με την τεχνητή νοημοσύνη και πολλά από αυτά τα θέματα έχουν ήδη διανύσει μακρύ δρόμο στα νομικά συστήματα. Πράγματι πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το θέμα και να δούμε καταρχήν τι είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Στο Ευρωπαϊκό Γραφείο για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα επισημάνθηκε ότι η τεχνητή νομοσύνη, τα big data και τα <clears throat> ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι οι θεμελιώδεις αρχές. Εγώ πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη συνυπολογίζεται και αυτό αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Κομισιόν. Αυτό που ενδιαφέρει είναι καταρχήν να βολιδοσκοπήσουμε, να δούμε ε, ποιες εξελίξεις ε, της τεχνητής νοημοσύνης παίζουν ρόλο για το νομικό σύστημα. Όλα αυτά σχετίζονται και με τη διαφάνεια. Οποτεδήποτε χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι στην τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς οφείλουμε να μεριμνήσουμε, να επικρατεί η διαφάνεια, έτσι ώστε πολίτες ε, να ξέρουμε κι εμείς ε, πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μας. Θεωρώ ότι όλα αυτά θα διδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συσταθεί ένα πλαίσιο έτσι ώστε να είναι δυνατόν να ε, χρησιμοποιείται η τεχνητή νομοσύνη για τη βελτίωση της ε, ανταγωνιστικότητας πολυεθνικών εταιριών. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να στηριχθούν οι επενδύσεις αυτών των εταιριών και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε νομοθεσία που να είναι ευέλικτη, η οποία αφενός ε, στηρίζει την καινοτομία, από την άλλη όμως ε, καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια το πώς πρέπει να προστατεύονται οι καταναλωτές ε, και πώς ακριβώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων αλλά και των ανθρώπων. Αυτό που έχει σημασία είναι η κείμενη νομοθεσία να εξετάζεται και κάτω από αυτό το πρίσμα. Μπορώ λοιπόν να φανταστώ ότι ε, σε κάποια σημεία θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω. Αυτό που ενδιαφέρει επίσης είναι το να δούμε λιγάκι τι γίνεται και με την οδηγία περί ανάληψη ευθυνών. Εκεί να συμπεριληφθούν ε, ορισμοί που προβλέπουν ε, τον περισμό αυτής της ευθύνης ή το θέμα της παραγραφής ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συνέστησε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων ακριβώς ε, για να τεθεί αυτό το θέμα της ανάληψης ευθυνών σε σχέση με την νέα τεχνολογία. Θεωρώ ότι η Προεδρία μας ε, θα περιμένει μέχρι να κατατεθούν συγκεκριμένα πορίσματα από την ομάδα των εμπειρογνωμόνων, αλλά βέβαια είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε πάνω σε αυτή τη βάση και πρέπει να σας πω και όλα αυτά θα μας απασχολήσουν ε, ουσιαστικά στο μέλλον. Φοβάμαι ότι η απάντησή μου ήταν λίγο μακροσκελής, αλλά ήθελα να απαντήσω λιγάκι διεξοδικά. Όσον αφορά το ερώτημα της ε, κυρίας Jones, δηλαδή το ερώτημα που αφορά στην ισότητα των δύο φίλων και στην σχετική οδηγία. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε κατά νου πρώτα απ' όλα ότι ε, στις, για τις επιχειρήσεις, ε, μάλλον στις επιχειρήσεις θα πρέπει να επικρατεί η ισότητα των δύο φύλων, γιατί αυτή είναι σημαντική για τις δυνατότητες ανάπτυξης που υπάρχουν για τις κοινωνίες μας. Το Δεκέμβρη του 2015 ε, τέθη το θέμα επιτάπητος και η ισότητα των δύο φύλων αντιμετωπίστηκε ως πρώτη προτεραιότητα για την επόμενη Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει επίσης ότι ακριβώς αυτή η πρόταση οδηγίας ε, πρέπει απαραίτητα να εξεταστεί περαιτέρω. Ε, η ε, επόμενη πρόεδρο της Επιτροπής έχει ήδη πει ότι θα ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Εμείς ως Φινλανδική Προεδρία θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να μεριμνήσουμε κι εμείς να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτή την κατεύθυνση. Πολύ ωραία. Ο κύριος Λεμπρετόν ε, για την επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Καλησπέρα, Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε τις προτεραιότητες της Φινλανδικής Προεδρίας και θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση για μία από τις προτεραιότητες που μας παρουσιάσατε, δηλαδή ε, καλύτερη τήρηση του κράτους δικαίου είναι ένα επίκαιρο ζήτημα γιατί στις 8 Απριλίου του 2019 η Επιτροπή κατέγραψε μία πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών που αφορούσε ακριβώς ε, την, ε, τον σεβασμό του κράτους δικαίου. Και εδώ έχουμε δύο διαφορετικές στάσεις. Είτε προωθούμε ένα σύστημα κυρώσεων, είτε, και αυτή είναι η δική μου προσωπική θέση, ενθαρρύνουμε ένα σύστημα διαλόγου και συνεργασίας. Υπάρχει το άρθρο 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που επιτρέπει την, ε, ε, τις κυρώσεις σε περιπτώσεις σφαλμάτων, ακόμη και κατάργηση του δικαιώματος ψήφου και αυτό έτυχε στην περίπτωση της Πολωνίας και Ουγγαρίας και υπάρχει και το, ο ετήσιος πίνακας αποτελεσμάτων για τη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας δίνει πολλές ενδείξεις που μας ενημερώνουν ε, για την κατάσταση αντεξαρτησίας ε, ε, των δικαστικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια θα είναι η κατεύθυνση που θα, προς την οποία θα προχωρήσετε. Ξέρω ότι πάρα πολλά γίνονται για να τονιστεί η πτυχή των κυρώσεων. Κάποια ψηφίσματα του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου του 2016 για ένα μηχανισμό ε, εποπτείας ε, των κυρώσεων. Ήμουν κατά του, του ψηφίσματος αυτού τότε, όπως είναι φυσιολογικό και δεν θα σας εκπλήξει. Και υπάρχει και μια ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Απριλίου του 2019 που εξηγεί πολύ σωστά ότι υπάρχουν τρεις πτυχές στην πρόθεση του κράτους δικαίου. Μια πρώτη πτυχή που είναι η πρόθεση όπως αποκαλείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι μια θετική πτυχή, δηλαδή εξηγεί τι είναι το κράτος δικαίου και μπορούμε να εμπνευστούμε από το έργο της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για να κατανοήσουμε τι είναι. Δεύτερη πτυχή είναι η πρόληψη δηλαδή διεξαγωγή διαλόγου και συνεργασίας με τις χώρες που αναγνωρίζουν τους κανόνες αυτούς και εδώ υπάρχει μία πρόταση που νομίζω σας έχει υποβληθεί, δεν ξέρω αν θα την ακολουθήσετε, δηλαδή να βελτιωθεί η ετήσια συζήτηση που γίνεται ήδη για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Συμβούλιο, για το κράτος δικαίου στο Συμβούλιο. Υπάρχει αυτή η διαδικασία, αλλά από ό,τι ξέρω δεν είναι πολύ αποτελεσματική και ορισμένε χώρε σα έχουν προτείνει να τη βελτιώσετε. Θα ήθελα λοιπόν να μα πείτε αν πρόκειται να κάνετε κάτι σχετικό. Και η τρίτη πτυχή που με φοβίζει προσωπικά είναι η πτυχή που αποκαλείται απάντηση στην ανακοίνωση της Επιτροπής και η απάντηση είναι οι κυρώσεις. Αυτή η απάντηση συνίσταται στο να, να επιβάλλονται ε, οικονομικές κυρώσεις στις χώρες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου. Θέλω λοιπόν να μας πείτε πώς βλέπετε αυτές τις πτυχές, αν θα προωθήσετε τη συνεργασία ή τις κυρώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία ευχαριστω η κυρια και μετά θα δώσουμε το λόγο στην Υπουργό να απαντήσει. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για το κράτος δικαίου υπό μια διαφορετική ε, πτυχή. Θα μιλήσω για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, και στις 24 ε, Ιουνίου μας υπενθύμησαν τα Ηνωμένα Έθνη την αλλαγή του κλίματος και όλες τις προσπάθειες για την εξάλληψη της φτώχειας, οι οποίες τίθενται σε κίνδυνο ακριβώς λόγω της κλιματικής αλλαγή και αυτό αποτελεί και ε, ε, παράγοντα για τον οποίο ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα θίγονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ευρώπη τα θύματα της κλιματικής αλλαγής και έχω συγκεκριμένο παράδειγμα αυτών που υπέβαλαν προσφυγή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ικανοποιούνται επαρκώς. Όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όλοι έχουν δικαίωμα ε, να υποβάλουν ε, τέτοιες ε, προσφυγές. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν ποια είναι τα σχέδιά σας για μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορούμε να δίνουμε βήμα στα θύματα, να δούμε πώς μπορούν να μην μένουν ατιμόρυτοι υπεύθυνοι για την κλιματική αλλαγή και τι σκοπεύετε να κάνετε από τη θέση σας για να οθήσετε τα κράτη-μέλη να δεσμευθούν υπέρ μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Thank Are you happy to answer να σας δώσω το λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Και οι δύο αναφέρατε τα θέματα σχετικά με το κράτος δικαίου. Και η απάντησή μου θα προσπαθήσει να τα καλύψει. Η Φινλανδική Προεδρία αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στο θέμα του κράτους δικαίου. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και βεβαίως θέλουμε να ενδυναμώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον μέσω αυτής της προσέγγισης. Η Φιλανδική Προεδρία πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό και στην πράξη να καταβάλουμε ό,τι είναι δυνατόν σε κάθε κράτος μέλος χωριστά, ούτως ώστε να τηρούνται σε ίσο βαθμό οι κανόνες του κράτους δικαίου είναι ένα κεντρικό θέμα για την Φινλανδική Προεδρία. Διότι τελικά πρόκειται για τις κοινέ μας αξίες και την ενίσχυσή τους και η τήρηση του κράτους δικαίου είναι βασική προτεραιότητα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι μία ισχυρή δέσμευση για τις κοινέ μας αξίες είναι πολύ σημαντική και θα ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινή μας προσπάθεια. Από πλευράς Φινλανδικής Προεδρίας ε, θα προσπαθήσουμε με θετικό ε, και ενεργό τρόπο να βρούμε λύσεις. Θα ενισχύσουμε τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, ούτως ώστε με ενεργό και αποτελεσματικό τρόπο να προωθήσουμε την τήρηση του κράτους δικαίου και των κοινών μας αξιών στα κράτη-μέλη. Θέλουμε ε, να ασχοληθούμε και με την πρόληψη των προβλημάτων, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να φτάσουμε σε κυρώσεις για να ενισχύσουμε ε, το κράτος δικαίου, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης ε, ήδη συζήτησαν το θέμα αυτό τον Ιούλιο στο άτυπο συμβούλιο στο Helsingfors και σε αυτή τη άτυπη σύνοδο των Υπουργών Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαμε ότι αυτό είναι θέμα ε, αρμοδιότητας των Υπουργών Δικαιοσύνης αλλά είναι πρώτη φορά που συζητήθηκε αυτό το θέμα του κράτους δικαίου ε, στο πλαίσιο Συμβουλίου Υπουργών. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο όπου θα καλύπτονται τα βασικά κριτήρια για το κράτος δικαίου και τίθεται το θέμα ε, του πώς θα ενισχύσουμε ε, το κράτος δικαίου κατά τα επόμενα έτη. Όπως σας είπα, ήδη ε, το συζητήσαμε στο Συμβούλιο Υπουργών τον Ιούλιο και είπαμε ότι θα υποστηρίξουμε τον σχετικό διάλογο. Και ε, κατά τη διάρκεια της Φινλανδικής Προεδρίας ε, θα κάνουμε διαπραγματεύσεις σε σχέση με έναν κανονισμό που θα μπορέσει να συσχετίσει περισσότερο τις αρχές του κράτους δικαίου αφενός και την χρήση ε, χρηματοδοτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφετέρου. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε ένα κανονισμό για το θέμα αυτό, ούτως ώστε να ενισχυθεί η αρχή του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τη συσχετίσουμε με την ε, χρηματοδότηση με ευρωπαϊκούς πόρους είναι μια βασική αρχή για τη δημοκρατία. Το κράτος δικαίου μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη διαφθορά, γιατί και η διαφθορά είναι ένας παράγων που θέτει σε κίνδυνο το κράτος δικαίου. Όσον αφορά την μακροπρόθεσμη το μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό προγραμματισμό και το πώς θα εφαρμόσουμε στην πράξη αυτά τα μέτρα, δεν έχουμε κατά νου να εφαρμόσουμε ένα μηχανισμό κυρώσεων, αλλά θέλουμε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορεί να αμυνθεί καλύτερα. Αυτό θα πρέπει να αρκεί για την ε, ενίσχυση του κράτους δικαίου και αποτελεί και τμήμα του προγράμματος της Φινλανδικής Προεδρίας. Τώρα για τα περιβαλλοντικά θέματα. Όντως η κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό θέμα για όλους ε, τους πολίτες του κόσμου, για ολόκληρο το πλανήτη. Και θα πρέπει με τις προσπάθειές μας να αναπτύξουμε μεθόδους και αποτελέσματα για την αποφυγή της κλιματικής αλλαγής. Και αυτό αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη Φιλανδική Προεδρία. Θα πρέπει από κοινού να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει η εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής Ε, κατανοώ απολύτω ε, τα μηνύματα της ε, βουλευτού που έλαβε το λόγο και μίλησε για την κλιματική αλλαγή. Και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα κάθε χώρα φέρει τη δική της ευθύνη για τα θέματα κλιματικής αλλαγής, αλλά και στη διεθνή κοινότητα θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να έχουμε στενότερη συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας, κυρία Υπουργέ, Κύριε Φόλκεν και κυρία Ομπρί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήρθατε σήμερα κοντά μας και θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή τύχη κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Γιατί πράγματι ζούμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή. Η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξελέγει οριακά και τώρα αυτό που επίκειται είναι η επιλογή των επιτρόπων. Ο κατάλογος ε, μοιάζει να είναι πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια φοβούμεθα ότι ε, κάποιοι επιτροποί ίσως ε, να μην ανταποκρίνονται στα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενδέχεται κάποιοι εξ αυτών να απορριφθούν από το Κοινοβούλιο. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σας ενθαρρύνω έτσι ώστε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων σας ως προεδρεύοντες να συμβάλλετε και εσείς ε, στο να έχουμε μία διαδικασία ε, που δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στο Κοινοβούλιο. Εντάξει, αυτό κατά κύριο λόγο είναι δουλειά της κυρίας Φόντα Λάιεν, αλλά σε τελική ανάλυση πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη, στην περίπτωση που υπάρξουν κάποιοι υποψήφοι που θα απορριφθούν από το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να τους αλλάξουν ε, και εκεί πρέπει να βοηθήσει η Προεδρία. Σας εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζω ε, πράγματι στο τέλος του έτους αυτού του τρέχοντος να έχουμε μία νέα επιτροπή. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε αυτά που ήδη ανέφερε η συνάδελφός μου, η κυρία Βάλτσμαν. Βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη και το ε, πώς θα προχωρήσουμε ως Ευρωπαίοι σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα κομβικό θέμα. Και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολούμεθα κυρίως με το θέμα της ανάληψης ευθυνών. Το ποιος φέρει την ευθύνη σε σχέση με την νοητή ε, τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα της ιδιοκτησίας εισαγωγικά. Για μας τους Ευρωπαίους έχει έρθει πια η στιγμή έτσι ώστε να καθορίσουμε προδιαγραφές σε διεθνές επίπεδο γιατί βλέπουμε ότι οι προδιαγραφές προκύπτουν εκεί όπου χρησιμοποιείται η τεχνολογία. Μπορεί κανείς να επικρίνει τον κανονισμό για την προστασία των ενδομένων αλλά πρέπει να αναγνωρίζει ότι εκείνο που κατόρθωσε είναι νωρί κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να ξυπνήσουμε λοιπόν όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και ελπίζω εσείς να συμβάλλετε προς αυτήν την κατεύθυνση. Το τελευταίο θέμα που θέλω να θίξω είναι το εξής. Εχθές, στο κατηάρκεια του δείπνου, είπατε ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ στην Προεδρία σας να είσαστε διαφανείς, να ενισχύσετε τη διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτό είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση ε, και πρέπει η δική σας η Προεδρία να δώσει το ε, καλό παράδειγμα. Ε, ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε, να δημοσιεύετε τις συναντήσεις, ε, όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται, αλλά στη δική σας την ιστοσελίδα, την εθνική. Και έτσι ε, θα αποκτήσετε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό που επίσης ενδιαφέρει είναι η έκθεση ε, αναχώρες, country by country reporting. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σκάνδαλα που είδαμε, Leaks, Panama Leaks, τα Panama Papers, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ήδη από το 2016 μια σχετική στρατηγική. Το 2017 στο Κοινοβούλιο εμείς καταλήξαμε στην ε, οριστική μας θέση και μεγαλύτερη διαφάνεια στο θέμα της φορολογίας, προφανώς αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά και ανάληψη ευθυνών και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να αποφύγουμε ή μάλλον να καταπολεμήσουμε την ε, φοροδιαφυγή αποτελεσματικά. Ε, ρωτώ, εσείς ως Προεδρία προτίθεστε να προχωρήσετε περαιτέρω σε επίπεδο Συμβουλίου όσον αφορά τις εκθέσεις αναχώρες και θεωρώ ότι τον τρόπο αυτό θα προσθέσετε στη διαφάνεια. Το εύχομαι. Και σας εύχομαι επίσης καλή επιτυχία ε, γιατί η φάση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι χρειάζεστε τις ευχές για καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Με κύριο Μπρι. Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Δεν συντονιστήκαμε, αλλά θα μπω ακριβώς στο θέμα που έθιξε και ο συνάδελφος και θα συνεχίσω να σας ρωτάω και εγώ για την αναχώρα έκθεση. Στην παρουσίασή σας το αναφέρατε και χαίρομαι γι' αυτό. Όμως σήμερα γνωρίζουμε ότι ο φάκελος ε, πάνω στον οποίο τσακωθήκαμε περισσότερο στην προηγούμενη θητεία και κινδυνεύουμε να μην προχωρήσουμε γιατί υπάρχουν διάφορες πολυεθνικές ε, που δεν το θέλουν. Με αυτή την δημοσίευση ε, των καταχώρα εκθέσεων θα γνωρίζουμε την πραγματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο και εκτός, γιατί και αυτό ήταν που συζητήθηκε στην προηγούμενη θητεία και το τι πληρώνουν από φόρους. Οι διατάξεις υπάρχουν ήδη στην οδηγία ΣΕΡΔΕ 4. Εγώ στην Oxfam, για παράδειγμα, έχουμε αναλύσει τα δεδομένα και ξέρουμε ότι είναι πολύ χρήσιμα να τα έχουμε αυτά τα τραπεζικά δεδομένα. Μπορεί να μην είναι η πανάκια για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή, αλλά σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε την φοροποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Οπότε ε, χαίρομαι και θα χαιρόμουν ακόμα περισσότερο αν μέσα στους επόμενους έξι μήνες μπορέσουμε να προχωρήσουμε το φάκελο αυτό. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με κάτι το οποίο δεν θίξατε καθόλου. Εδώ είμαστε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και υπάρχει ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετούς ε, βουλευτές που έχει να κάνει με την εποπτεία και την προστασία. Υπάρχει ατιμορρησία νομικά απέναντι σε διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες ε, προμηθευόμενες τα προϊόντα τους ε, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και έχουμε πάρα πολλά σκάνδαλα τέτοια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαιτία του νομικού κενού. Είμαι Γαλλίδα και υπάρχει μια τέτοια νομοθεσία στη Γαλλία η οποία έδειξε ότι είναι πολύ σημαντικό να διώκεται νομικά η ευθύνη αυτή εφόσον παραβιάζεται και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη δυνατότητα, για την αποφασιστικότητά σας, την πολιτική σας βούληση, εν πάση περιπτώσει, της Φιλανδίας να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση και να καταλήξει σε μια πρόταση την οποία εμείς περιμένουμε και είναι κρίμα που δεν είναι κοινοβουλευτική αυτή η πρωτοβουλία, τι να κάνουμε, αυτό είναι άλλη συζήτηση, αλλά να έχουμε από εσά μια πρόταση θα την κάνει φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς να την στηρίξετε, γιατί προς το παρόν δεν την βλέπω στις προτεραιότητες της Φιλανδικής ε, Προεδρίας. Να απαντήσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει το θέμα της διαφάνειας. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για τις εξαιρετικές ερωτήσεις που μας θέσατε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ενθαρρυντικά λόγια τα οποία απευθύνονται προς εμένα. Όσον αφορά τη διαφάνεια, υπάρχει το στρατηγικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2024 και εδώ έχουμε την εξέλιξη των μεθόδων εργασίας του Συμβουλίου με κατεύθυνση τη διαφάνεια. Προσπαθούμε να δείξουμε ότι με μεγαλύτερη διαφάνεια θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στραφεί περισσότερο στους πολίτες και να κερδίσει και την εμπιστοσύνη των πολιτών αυτό είναι κάτι που θέλουμε να προωθήσουμε ως Προεδρία του Συμβουλίου με κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου, παραδείγματο χάρη, περισσότερες συνεδριάσεις θα είναι δημόσιες. Θα δίνουμε περισσότερες πληροφορίες για τις διάφορες συναντήσεις του Συμβουλίου. και θα δίνουμε πληροφορίες και για σχέσεις με ε, ομάδες πιέσεων ε, και λόμπι. Θα προσπαθήσουμε και στα νομοθετικά κείμενα να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Και η πρόσβαση σε πληροφορίες και η δημοσιότητα θα δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε καλύτερα την παραπληροφόρηση τα μέσα ενημέρωσης, ε, το Twitter πολύ συχνά διαχέουν εσφαλμένες πληροφορίες και αυτή την παραπληροφόρηση μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη δημοσιοποίηση των δικών μας δραστηριοτήτων. Μετά, για την υποβολή εκθέσεων αναχώρα. σχετικά με την, τα ποσά φόρων τα οποία καταβάλλονται σε κάθε χώρα. Θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τις ενέργειες στον τομέα αυτό δεν είναι μόνο ότι η νομική βάση πολλές φορές είναι διαφορετική και δυσκολεύει την κατάσταση. Θα προσπαθήσουμε όμως να εξετάσουμε το θέμα πολύ προσεκτικά και ε, να προωθήσουμε τις ε, δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτό το θέμα. είναι σημαντικό για τα θέματα φορολογίας, γιατί όταν δημοσιοποιούνται πληροφορίες ε, μπορούμε να υποχρεώσουμε τις επιχειρήσεις πιο εύκολα ε, να αναλάβουν ε, τις ευθύνες τους και να υπάρχει πιο δίκαιη φορολόγηση. Αυτό είναι σημαντικό για την κυβέρνηση της Φινλανδίας. Είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και που θέλουμε να προωθήσουμε. Και τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν σήμερα αποτελούν προτεραιότητές μας. μπορούμε ε, και να συνεχίσουμε τη συζήτηση του θέματος, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό και να παράσχουμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα, για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και για τις δραστηριότητες ε, εταιριών, Ήδη υπάρχουν ε, δικαστικές ε, διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν είναι άμεσα ε, στις δικές μου αρμοδιότητες το θέμα αυτό, αλλά σίγουρα θα προωθήσω το θέμα αυτό στους αρμόδιους συναδέλφους. Είναι πολύπλοκα θέματα τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Um, Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχω άλλες τέσσερις ερωτήσεις. Ας ακούσουμε τις δύο πρώτες. Κυρία Μέρκερ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω εάν υπάρχει διερμηνία στα δανέζικα στη γλώσσα μου, οπότε επανέρχομαι στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην Επιτροπή μας. Στην ομάδα μας, στην ομάδα Renew Europe, ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα την έμφαση την οποία δίδεται στα θέματα εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα και στο κράτος δικαίου Και αυτό είναι σημαντικό για να μπορέσουν να έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτες της Ευρώπης στα θεσμικά όργανα και στα εθνικά θεσμικά όργανα. Κατά τα επόμενα πέντε χρόνια θα πρέπει να ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι εμείς ως θεσμικά όργανα εργαζόμαστε υπέρ των πολιτών και όχι υπέρ κάποιων σκιωδών συμφερόντων. Κάποια θέματα, κάποια νομοθετικά θέματα έχουν παγώσει στο Συμβούλιο. Ένα από αυτά είναι για τους whistleblowers, για τους κοινοποιούντες πληροφορίες και θα ήθελα να μας πείτε αν προτίθεστε να το προωθήσετε, γιατί θέλουμε να προστατεύονται τα άτομα τα οποία εφιστούν την προσοχή σε ε, παρατυπίες και θα θέλαμε να ε, ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Όπως και για το θέμα της υποβολής εκθέσεων αναχώρα και της ε, ιτερικής ευθύνης. Χαίρομαι για αυτά που είπατε για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, γιατί είναι πολύ σημαντικό να είναι στεναρή η θέση μας επί του θέματος και η νομοθεσία που έχει θεσπιστεί θα πρέπει να υλοποιείται. η ευθύνη των κρατών μελών ε, στο να εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία θα είναι ε, κομμάτι των προτεραιοτήτων της Προεδρίας σας. Υπάρχουν κάποιες ε, περιπτώσεις ξεπλήματος χρήματος όπου η χώρα μου, η Δανία, δεν μπορούσε να δει ότι κάποια τράπεζα στη Δανία είχε τέτοιες δραστηριότητες παράνομες, ε, ενδεχομένως και μέσω της θηγατρικής της, στην Εστονία. Πώς μπορούμε να έχουμε ε, αρκετά ισχυρό πλαίσιο για να μπορούμε ε, να παρακολουθούμε τέτοια περιστατικά, όπως θα το επιθυμούσαν οι νομοθέτες οι οποίοι έχουν θεσπίσει, το, θεσπίσει το, σχετικό, τη σχετική νομοθεσία. Η Νέα Επιτροπή νομίζω θα συνεχίσει το πρόγραμμα που έχει ήδη ξεκινήσει στην προηγούμενη θητεία για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα ήθελα να ακούσω και από εσά ποια είναι τα σχέδιά σα για το πώ μπορούμε να κερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών και για τι αποφάσει οι οποίε λαμβάνονται και για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών σε θέματα τεχνητή νοημοσύνη. Ευχαριστώ. Η κυρία Πόλτερ είναι η επόμενη ομιλητρία. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία κατά τη Φιλανδική Προεδρία. Δύο ερωτήσεις. Μιλήσατε για την διαφάνεια στα θεσμικά μας όργανα, που είναι πολύ σημαντικό αλλά πολύ σημαντικό είναι και η διαφάνεια για τις εταιρείε. Ανέφερε ο συνάδελφος και άλλοι συνάδελφοι την υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Ένα άλλο θέμα είναι η λογοδοσία των εταιριών, το τι ε, δηλώνουν οι εταιρείε και πώς το δηλώνουν. Έχει υλοποιηθεί η οδηγία για την υποβολή ε, ε, εκθέσεων, αλλά υλοποιείται με διαφορετικό τρόπο από κάθε εταιρεία και στο μεταξύ η οδηγία δεν πληρεί τους στόχους για τους οποίους θεσπίστηκε. Έχω ακούσει ότι ε, μπορεί να υπάρξει κάποια αναθεώρηση της οδηγίας από την Επιτροπή. Το Συμβούλιο προετοιμάζεται για κάτι τέτοιο. Θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία το Συμβούλιο πριν από κάποια σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα θέλαμε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά η ερώτησή μου καταρχήν είναι αν η Προεδρία σας σκοπεύει να κάνει κάτι κατά τους προσεχείς μήνες. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά τις συλλογικές προσφυγές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει θέση από αυτού. Το ε, Συμβούλιο είναι έτοιμο ε, Είναι... Το Συμβούλιο δεν έχει προς το παρόν κάτι ε, σχετικό και αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια πολιτών στην Ευρώπη δεν έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και μπορεί να υπάρχει ένα όχημα της Volkswagen που ρηπαίνει την ατμόσφαιρα και να μην μπορούν να αντιδράσουν οι πολίτες, δεν μπορούν συλλογικά να εξασφαλίσουν δικαιοσύνη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι αν η Προεδρία σας θα ξεμπλοκάρει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Tack Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τους ε, δυο σας για τις πάρα πολύ καλές ε, ερωτήσεις. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσω με την Κάρεν. Δυστυχώς και τα δικά μου τα δανέζικα φτωχά είναι, γι' αυτό θα προτιμήσω να μιλήσω σουηδικά, να συνεχίσω στα σουηδικά. Ίσως λοιπόν για την οδηγία σχετικά με τους ε, καταγγέλλοντες ε, μπορούμε να πούμε τα εξής. Ε, το θέμα εξετάστηκε ήδη κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας και επ' αυτού επιτεύχθηκε κάποια συμφωνία επί της οδηγίας και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Υπήρξαν περιπτώσεις κατάχρησης όπου γνωστοποιήθηκαν κάποια στοιχεία για κάποιους ανθρώπους και ε, οι άνθρωποι αυτοί έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι οποτεδήποτε γίνεται κάποια αναφορά και χρήση πληροφοριών, θα πρέπει να υπάρχει και σιγουριά, ασφάλεια. Η προστασία των καταγγελόντων ε, πρέπει να ενισχυθεί. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Ε, πράγματι μας ενδιαφέρει ο πιο θεμητός ανταγωνισμός και είναι απόλυτα σαφές ότι θέλουμε να υπάρχουν ίσοι όροι, δίκαιοι όροι οι δικοί μας, οι, οι συμπολίτες μας πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο και ως εκ τούτου στο σημείο αυτό ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και να ευχαριστώ ιδιαίτερα αυτήν την Επιτροπή γιατί ε, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκείνο το οποίο κατά κύριο λόγο έθιξε αυτά τα θέματα. Αυτή η οδηγία πρέπει επιτέλους να εγκριθεί και να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο. Εμείς ως Φινλανδική Προεδρία θα συνεχίσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Τόσο, τώρα, όσον αφορά στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ε, κοινοποίησε μία οδηγία και σε αυτήν μια έκθεση μάλλον και σε αυτή την έκθεση αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη και οι αρμόδιοι φορείς πρέπει οπωσδήποτε να ε, στηριχθούν στον αγώνα τους στην καταπολέμηση αυτών των ε, δραστηριοτήτων γιατί όλα αυτά αναμφίβολα συνδέονται και με τρομοκρατικές ενέργειες. Τώρα πλέον η νομοθεσία για την νομοποίηση αυτών των παράνομων εισόδων ε, η νομοθεσία είναι πολύ πιο αυστηρή αλλά σε εθνικό επίπεδο εδώ ε, δεν εφαρμόζονται πολλά στοιχεία της νομοθεσίας. Εκεί πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί να εφαρμόζονται. Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι κανόνες είναι αποτελεσματική, αλλά θα πρέπει και να εφαρμόζονται σωστά. Και σε όλα τα κράτη θα πρέπει το θέμα να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και από αυτού του θέματος πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με άλλους ε, διεθνείς οργανισμούς, ε, παραδείγματος χάρη με την Task Force ε, της, που ονομάζεται Financial Action και δραστηριοποιείται υπό την αιγίδα του ΟΣΑ. Το θέμα λοιπόν της ε, καταπολέμησης της ε, νομοποίησης παράνομων εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν είναι σωστό να υπάρχει αυτή η δραστηριότητα. Οι αρμόδιοι φορείς ε, οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το όλο θέμα και νομίζω ότι και αυτό, όπως και το θέμα των ε, καταγγελόντων, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον, οποτεδήποτε θα τεθεί επιτάπητος ε, το θέμα των δραστηριοτήτων ε, που είναι παράνομες και ως εκ τούτου πρέπει να εκλείπουν. Τώρα, όσον αφορά ε, στις ε, συλλογικές ε, προσφυγές. Τώρα, εδώ με τη συνάδελφό μου τα λέμε μισά φιλανδικά, μισά σουηδικά. Ε, θίξατε το θέμα των συλλογικών προσφυγών. Ε, για μας ε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ακριβώς όπως τονίστηκε από την κυρία Ευρωβουλευτή. Πράγματι πρέπει να ενισχυθεί η θέση των καταναλωτών στην κοινή αγορά. Και αυτό το θέμα, το θέμα των συλλογικών προσφυγών, είναι ένα θέμα καθοριστικής σημασίας ε, να υπάρχει μια νέα συμφωνία για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Βεβαίως, ε, όλα αυτά πρέπει και να εφαρμόζονται στην πράξη για να ενισχυθεί η θέση των ε, καταναλωτών και για να υπάρχει η δυνατότητα να προστατεύονται και οι επιχειρήσεις από το ενδεχόμενο κατάχρησης τέτοιου είδους ε, μαζικών ε, προσφυγών. Εμείς, ε, κατά τη διάρκεια της Φινλανδικής Προεδρίας, έχουμε αποφασίσει το φθινόπωρο να θεσπιστεί μια οδηγία επί του θέματος και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ οι δύο τελευταίες ερωτήσεις. Τώρα κύριε Χαουτάλα πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε. Με εκπλήσει το καλωσόρισμα στην Φιλανδική Προεδρία. Ε, μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη προεδρία που δίνει τόσο μεγάλη σημασία στο κράτος ε, δικαίου. Και αυτό είναι αξιοσημείωτο πραγματικά. Τώρα, θέλω να σας υπενθυμίσω ένα πρόγραμμα που ίσως να το γνωρίζετε. Εδώ και πολλά χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχει προωθήσει και έχει προτείνει νομοθετική πρόταση για διοικητικές διαδικασίες από πλευρά κράτου δικαίου, αυτή η οργάνωση που τόσο πολύ έχει προχωρήσει και έχει οριμάσει, δεν διαθέτει τις διοικητικές διαδικασίες. Εμείς ε, λέμε ότι θέλουμε μια ανοιχτή ευρωπαϊκή δίκηση κτλ. Έχουμε το άρθρο 298 της συνθήκης της Λισαβόνας, αλλά είναι η μόνη νομική βάση η οποία δεν οδήγησε σε νομοθεσία τελικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν θα μπορούσε να βασίσει τις ελπίδες του στη Φιλανδική Προεδρία, η οποία αντιλαμβάνεται τι σημαίνει χρηστή δίκηση και καλή διοικητική αντιμετώπιση, που για μας είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση εσείς ως Προεδρία να θελήσετε να το θέσετε αυτό το ζήτημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί τελικά πρέπει κάτι να κάνουμε για να προχωρήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντάει λέγοντας «Ε, έχουμε τον κώδικα δεντολογίας μας για τις καλές διοικητικές πρακτικές. Ναι, αλλά ίσως δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουμε νομοθεσία δεσμευτική και ότι έχουμε 50 διαφορετικά υπηρεσίες, οργανισμούς ε, κλπ που εφαρμόζουν διαφορετικές διοικητικές πρακτικές. Και αυτό είναι ιδιαίτερα περίπλοκο για τον ε, πολίτη Συνεπώς, τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε από τη Φιλανδία από αυτού. Και όσον αφορά επίσης το κράτος δικαίου, αναφερθήκατε συχνά στην διαφάνεια. Ε, τον Απρίλιο κάπου 100 ευρωβουλευτές έστειλαν επιστολή στη Φιλανδική Προεδρία ζητώντα μέτρα υπέρ της διαφάνειας. Δύο πράγματα έχω να πω εδώ. Ζητήσαμε από τη Φιλανδική Προεδρία να διασφαλίσει ότι τα πρακτικά των ε, ομάδων εργασίας θα δημοσιοποιούνται με τα ονόματα των κρατών μελών και θα θέλαμε η νομοθεσία να το υποχρεώνει αυτό. Μπορείτε να το κοιτάξετε αυτό. Επίσης υπογραμμίσαμε ότι τελικά η Προεδρία δεν έχει κανόνες και ξέρω ότι ο συνήγορος του πολίτη, ο Όμπουτσμαν, ο Ευρωπαίος, το έχει θίξει, εσείς το έχετε κοιτάξει καθόλου και πώς θα αντιδράσετε. Τέλος, ίσως να το διαπιστώσατε ότι όλοι ενδιαφερόμαστε για τη λογοδοσία από, όλα, από όλες τις πλευρές του φάσματος και έχει αναφερθεί κάτι για πλαίσιο ευρωπαϊκό, για ευρωπαϊκά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε μήπως πράγματι ήρθε η ώρα να τεθεί το ζήτημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι δεν είναι αυτό καθ' αυτό δικιά σας αρμοδιότητα, αλλά υπάρχουν σημαντικές πτυχές που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη των θυμάτων. Και αυτό είναι δική σας αρμοδιότητα. Οπότε μήπως θα θέλατε να δράσετε και προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να έχουμε σύντομα από την Επιτροπή μια νομοθετική πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λαγκατίνσκι έχει την τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Αφού μιλάνε όλη τη γλώσσα τους, θα μιλήσω και εγώ γερμανικά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ που ήρθατε εδώ ε, μιλήσατε για το κράτος δικαίου. Αυτό είναι το σημείο κίνηση της συζήτησής μας και έχουμε το έγγραφο της ε, Κομισιόν για το θέμα του κράτους δικαίου. Και ένα θέμα που υπάρχει σε αυτή τη συμφωνία είναι η προστασία της κοινωνίας των πολιτών. Εδώ λοιπόν ε, στη δική μας την Επιτροπή ένας τρόπος για να υπάρχει αυτή η προστασία είναι το εταιρικό δίκαιο ή το δίκαιο των ε, ε, ενώσεων, των συνασπισμών. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενοποιημένο δίκαιο και δεν έχουμε και ενοποιημένο δίκαιο για κοινοφελείς ε, δραστηριότητες και κοινοφελείς οργανισμούς. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί ξέρετε κάτι, σε κάποιες χώρες, σε κάποιες ενώσεις Κάποιες, κάποιοι συνασπισμοί ε, αναγκάζονται, είναι υποχρεωμένοι μάλλον οι οργανισμοί αυτοί, να δηλώνουν ε, τις χρηματοδοτήσεις που έχουν από το εξωτερικό. Σε άλλες πάλι χώρες υπάρχουν ε, ε που δεν αναγνωρίζονται ως κοινοφελείς οργανισμοί, μάλλον ως οργανισμοί που προσφέρουν στο κοινό καλό, απλά γιατί δραστηριοποιούνται πολιτικά. Άρα δηλαδή πρέπει να ενοποιηθεί κάπως η κατάσταση. Πρέπει να σας πω όμως ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια νέα προσέγγιση τόσο για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όσο και για το δίκαιο που διέπει ενώσεις, συνασπισμούς, οργανισμούς. Πιστεύετε εσείς ότι έχει φτάσει πια η χρονική στιγμή έτσι ώστε να γίνει κάτι συγκεκριμένο για την κοινωνία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Bra, tack för dessa frågor. Ναι, σας ευχαριστώ και για αυτές τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Χάουταλα. Μίλησα για το διοικητικό δίκαιο. Εκτός ε, πρακτικών, θέλω να πω ότι γνωριζόμαστε εδώ και χρόνια, κάποτε υπήρξαμε και μέλη τη ίδιας με την κυρία Χάουταλα. Όσον αφορά λοιπόν ε, το διοικητικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα θέλουμε ε, μια σωστή διοίκηση και επομένως το διοικητικό δίκαιο παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν υπάρχει η νομική βάση αυτή τη στιγμή για τέτοιου είδους διοικητικό δίκαιο, αλλά από δική μου πλευράς θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για τις εργασίες που έχει ήδη ε, κάνει για να προωθήσει αυτό το θέμα. Καταλαβαίνω ότι και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει μεγάλη σημασία το θέμα. Ας περιμένουμε τώρα ε, εάν ε, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει κάτι σε σχέση με το άρθρο 298. Νομίζω ότι εδώ και πάνω από 10 χρόνια υπάρχει κάποια βάση την οποία μπορεί να επαυξήσει η Επιτροπή. Η καλή διοίκηση η χρηστή διοίκηση ε, θα ενισχύσει και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ε, και αυτό ε, άπτεται και του θέματος της διαφθοράς. Θα το συζητήσουμε τον Οκτώβριο και είναι επίσης πολύ σημαντικό θέμα. και είναι ξεκάθαρο ότι συσχετίζονται αυτά τα θέματα. Η προώθηση της χρηστής διοίκησης συμβαδίζει με την καλύτερη νομοθεσία το διοικητικό δίκαιο, οι κανόνες για την χρηστή διοίκηση είναι κάτι που θέλουμε να προωθήσουμε, θέλοντας να προωθήσουμε και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Θέλουμε να δούμε πώς ε, μπορούμε να συσχετίσουμε την καλή διοίκηση με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και την συνάντηση του Οκτωβρίου θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να συσχετίσουμε τα δύο αυτά θέματα. Για το θέμα του sponsoring που με ρωτήσατε. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω για το ποια είναι τα θέματα τα οποία προωθεί η Φινλανδική Προεδρία. και για το sponsoring στα πλαίσια της Φινλανδικής Προεδρίας. Δεν ξέρω αν ε, αναλαμβάνουν χορηγίες κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες. Ε, ξέρω ότι στη Φινλανδία υπάρχει κάποια ε, ε, εταιρεία αυτοκινήτων που προσφέρει αυτοκίνητα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει και αντίστοιχα εταιρεία ποδηλάτων ή κάτι τέτοιο που θα μπορούσε να αναλάβει σχετικέ χορηγίες. Για την κοινωνία των πολιτών, ε, θέλω να πω ότι είναι πυλώνας της δημοκρατίας. Θέλουμε να συμμετέχουν οι πολίτες Και αυτό άμεσα έχει σχέση και με το κράτος δικαίου. Τα κράτη-μέλη πρέπει να προωθούν ε, συλλόγους πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί μια δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ενεργό συμμετοχή των πολιτών, χωρίς μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτά έχω να πω επί του θέματος, γιατί έμεσα και αυτό συνδέεται με το πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί το χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο τίθεται, η χρηματοδότηση όλων αυτών των θεμάτων, είναι ένα εργαλείο για την ενίσχυση της συμμετοχής, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών. τα δικαιώματα και οι αξίες των πολιτών είναι ένας από τους τομείς που προωθούνται μέσω του ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Τα καταφέρατε πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και είναι εντυπωσιακό που απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με θέματα όπως είναι το κλίμα, η φοροαποφυγή, η τεχνητή νοημοσύνη. Ένα πολύ ευρύ ερωτήσεων δηλαδή. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ και χαιρόμαστε που επικεντρώνεστε στο κράτος δικαίου. Θα συνεργαστούμε μαζί σας ε, για αυτό το ζήτημα και σίγουρα θέλουμε να ξέρουμε περισσότερα για τα συγκεκριμένα κριτήρια όσον αφορά τις διαδικασίες προσφυγής επί παραβάση. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για τις απαντήσεις σας. Ευχόμαστε όλοι στην Προεδρία σας κάθε επιτυχία. Είναι 4 και 20. 4,5 θα συνεχίσουμε. 10 λεπτά διακοπή και 4,5 θα συνεχίσουμε. Η Υπουργό, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και σα ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ για τι ερωτήσει σα. Και εγώ σα εύχομαι ότι καλύτερο η δουλειά που κάνετε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντική. Καλή επιτυχία λοιπόν και σε εσά και προσβλέπω και εγώ στην καλή μας συνεργασία. Um, λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε και πάλι. Η ώρα είναι 4.30. Έχουμε τους δύο υποψηφίους τώρα να εξετάσουμε για τη θέση του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Διονοτική Ιδιοκτησία. Ήρθαν, θα κάνουν κάποια σύντομη δήλωση Και πρέπει να σας πω ότι πριν καταλήξει το Συμβούλιο, η Επιτροπή μας έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει τους υποψηφίους που βρίσκονται στη short list και να τους υποβάλει ερωτήσεις. Οπότε σήμερα προσκαλέσαμε δύο υποψηφίους που έχουν προταθεί στο Συμβούλιο μετά από την συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΓΙΠΟ της 4ης Ιουνίου. Έχουμε τον Αντρέα Τικάρλο, και την Κάι Χάρμαντ. Καλώς ήρθατε και οι δύο. Έχουμε κυκλοφορήσει τις υποψηφιότητές σας, τα βιογραφικά σας, έχει φροντίσει η γραμματεία δηλαδή γι' αυτό. Τώρα έχετε ενημερωθεί ότι έχετε 10 λεπτά για να κάνετε κάποια παρουσίαση και άλλα 10 λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Ντικάρλιο λοιπόν. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και οι δύο εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Αύριο θα είναι 25 χρόνια που υπάρχει το γραφείο αυτό, το Ευρωπαϊκό Διανοητική Ιδιοκτησία. Έχει μεγαλώσει, έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και ιδιαίτερα δημοφιλές. Πάνω από 2 εκατομμύρια σήματα και 1,3 εκατομμύρια ε, σχέδια έχουν υποβληθεί από ολόκληρο τον κόσμο. Και όλο και περισσότερες αρμοδιότητες αναλαμβάνει όσον αφορά τη διεθνή σκηνή που έχουν να κάνουν και με θέματα συμμόρφωσης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης των πολιτών αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο όργανο αυτό προκειμένου να αποφέρει καρπούς. Και πάντα η βασική μας αρχή, όπως και πρόσφατα είπε το λεκτικό συνέδριο, είναι ότι το γραφείο μας πρέπει να είναι σε θέση να φροντίζει για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Σε στενή συνεργασία λοιπόν με τις Εθνικές Υπηρεσίες Δυνοτικής Ιδιοκτησίας στις χώρες μέλη και με τη βοήθεια του προσωπικού η υπηρεσία μας σίγουρα έχει στεφθεί με επιτυχία. Χαίρομαι λοιπόν και είμαι περήφανος για την δικιά μου συνεισφορά στην επιτυχία αυτή μέσω της πραγματογνωμοσύνης μου και του ενθουσιασμού μου. Σήμερα λοιπόν ξέρουμε όμως ότι δεν μπορούμε να επαναπτυχθούμε, ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε ώστε να μπορεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ιδιωτικής Ιδιοκτησίας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενισχυθεί η προστασία της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Ιδιοκτησίας και να υπάρχει και εύκολα πρόσβαση όλων στο γραφείο μας. Έχοντας υπόψη μας αυτά, υπάρχει ένα πρώτο στρατηγικό σχέδιο για τα επόμενα ε, πέντε χρόνια, το οποίο υποβλήθηκε και συζητήθηκε στην ε, τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και στη συνάντηση αυτή, εκπρόσωποι χωρών ε, μελών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασαν τη στήριξή τους στο σχέδιο αυτό. Και υπήρξε και ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μάλλον θα υπάρξει τον επόμενο μήνα. Θέλω τώρα εδώ να υπογραμμίσω ποια είναι τα βασικά στοιχεία του σχεδίου αυτού και πού μπορώ εγώ με τη δικιά μου εμπειρία να βοηθήσω σε αυτό. Ενώ οι αρμοδιότητες του Βεκού Γραφείου Διονετικής Ιδιοκτησίας έχουν επεκταθεί τελευταία, αλλά πρόκειται κυρίως για την ε, συνέχεια που θα δώσουμε και πώς θα ενισχύσουμε με το στρατηγικό αυτό σχέδιο τον ε, έλεγχο που έχουμε στη διανοητική αυτή ιδιοκτησία. Θέλουμε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες και να βελτιώσουμε την ποιότητα, την ε, συνέπεια και την αποτελεσματικότητα. Πρέπει οι χρήστες να μπορούν να συνεχίσουν να μας εμβουλεύονται. Η συνεργασία επίσης με περιφερειακά και εθνικά γραφεία διονετικής ιδιοκτησία, χρειάζονται κάποιον εξυγχρονισμό, έτσι ώστε να υπάρχει προστασία με το λιγότερο δυνατόν κόστος. Με το πρόγραμμα αυτό το νέο θα φροντίσουμε να βοηθήσουμε τους χρήστες, να το στηρίζουμε και να υπάρξει και επένδυση και σε νέους τομείς. Και ένα τέτοιο τομέα είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπω είπε και η πρόεδρος Φοντερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωπαϊκέ μικρομεσαίες επιχειρήσει είναι καινοτόμε και είναι η σπονδυλική στήλη τη οικονομία μα. Προσβλέποντα λοιπόν στο μέλλον, πρέπει η βιομηχανική πολιτική μας να βασιστεί στην ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτε του γραφείου μας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον ένα copyright σε εμά έχουν πολύ περισσότερε πιθανότητες να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν περισσότερο. Όμως, λιγότερο από 10% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, καταθέτουν και καταχωρούν σε εμά κάποια καινοτομία για να προστατευτεί. Συνεπώς εμείς πρέπει να εργαστούμε με τα Εθνικά Γραφεία διανοητική Ιδιοκτησίας για να μπορέσουμε να παίξουμε μεγαλύτερο ρόλο βοηθώντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην καινοτομία και να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ακόμα καλύτερα την, ε, τις διάφορες εφευρέσεις τους. Έτσι λοιπόν πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες σε συντονισμό βέβαια με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και σε στήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι καινοτόμε όμω μικρομεσαίε επιχειρήσει, όπω και επιχειρήσει γενικά, χρειάζονται προστασία απέναντι στον αθέμητο ανταγωνισμό. Και εδώ οι διαδικασίε επί είναι πολύ σημαντικέ. Για να αντιμετωπιστούν τα πλαστά προϊόντα, οι αντιγραφές, η πειρατεία που κοστίζει πάρα πολλά χρήματα ε, και πάνω από 50.000 θέσεις απασχόλησης. Τα τελευταία χρόνια η υπηρεσία μας μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήου για τις παραβιάσεις έχει συνεισφέρει σε καλύτερο συντονισμό με την αστυνομία, τα τελωνία, εισαγγελίε και δικαστές. Έτσι λοιπόν τώρα πρέπει να λυθούν πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να επωφεληθούμε από αυτόν τον συντονισμό, ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να βασιστούν σε αποτελεσματικές διαδικασίες, όχι μόνο για να, κατηχωρούν, να κατοχωρούν την ιδιοκτησία τους, την πραγματική ιδιοκτησία τους, αλλά και για να προστατεύεται αυτή και στη συνέχεια. Συγχρόνως, χρειάζεται και κάποια εκστρατεία επικοινωνία σε συντονισμό με τις εθνικές αρχές, ώστε να ενημερωθούν κατάλληλα και οι καταναλωτές, οι οποίοι όλο και περισσότερο είναι εκτεθειμένοι σε προϊόντα που μπορεί να είναι και επικίνδυνα ή να μην είναι ασφαλή και από τα οποία υποφελείται το οργανωμένο έγκλημα. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία και με τα Υπουργεία Παιδείας των χωρών μελών. Τέλος, τεχνολογία. Η τεχνολογία ε, είναι αυτή που μπορεί να βοηθήσει τη στρατηγική μας στο μέλλον. Η τεχνητή νοημοσύνη τα μεγάλα δεδομένα, blockchain, είναι πράγματα τα οποία διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η υπηρεσία μας και επικοινωνεί με τους χρήστες. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή και φέτος και συνεργαζόμαστε με, τα περισσότερα, με τις περισσότερο καινοτόμες υπηρεσίες στον κόσμο. Θέλουμε τις καλύτερες προδιαγραφές και για το περιβάλλον και για τις προσφορές, ώστε να μπορεί να υπάρξει πλήρης ανάπτυξη. Μπορεί επίσης το γραφείο μας όμως να συνεισφέρει με την εμπειρία του να προσφέρει λύσεις σε άλλη τα μέχρι τώρα προβλήματα. Και αυτό γίνεται, για παράδειγμα, με την blockchain όσον αφορά τα πλαστά προϊόντα, σε συνεργασία με επιχειρήσεις ε, τεχνολογίας, με την αστυνομία, με τα τελωνία και έτσι θα αναπτυχθεί καλύτερα η υποδομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση ε, των ε, πλαστών προϊόντων. Αυτά τα χρόνια λοιπόν έχουν χρησιμεύσει για να καθοριστεί το μέλλον. Η θέση του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή έχει σαν στόχο ακριβώς τη στήριξη όλων αυτών ε, των σχεδίων. Ως μέλος της ε, Steering Επιτροπής ε, για το στρατηγικό αυτό σχέδιο έχω βοηθήσει στη διαμόρφωση του σχεδίου και έχω κερδίσει γνώση μέσα από την υπηρεσία. Είχα και ηγετικό ρόλο σε διάφορους τομείς όπως είναι η δίκηση, όπως είναι τα συστήματα καταχώρησης, οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες, συνεργασία με τις Εθνικές Υπηρεσίες Προστασίας Διανοητικής ε, Ιδιοκτησίας και Θέμη επίσης υπεύθυνο ως επικεφαλής ενός ε, προγράμματος από τα πιο σημαντικά για την τροποποίηση στον ε, τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Όλα αυτά απαιτούν διαχείριση και χρημάτων αλλά και προσωπικού, όπως επίσης και συνεργασία με το κοινό, με τους χρήστες και μέχρι τώρα έχω δείξει ότι μπορώ να έχω αποτελέσματα μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον και πολυπολιτισμικό, όπως είναι αυτό μέσα στο οποίο δρά το γραφείο μας. Μπορώ λοιπόν να διασφαλίσω ε, ότι θα προσφέρω τη γνώση μου, τη δυνατότητά μου να ηγηθώ και την εφαρμογή του νέου αυτού στρατηγικού σχεδίου. Βάσει των ε, καλών σχέσεων συνεργασίας που έχω επίσης με τον εκτελεστικό διευθυντή έχουμε μια κοινή αντίληψη για το μέλλον της υπηρεσίας και πιστεύω ότι συμπληρώνουμε ένα τον άλλον με τις εμπειρίες που έχουμε τώρα. Έπειτα θα είναι τιμή μου να βοηθήσω τον ε, εκτελεστικό διευθυντή να συνεχίσει, όπως και το γραφείο μας, στον δρόμο επιτυχίας στον οποίο βρίσκεται, με τη βοήθεια βέβαια του προσωπικού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much indeed. Um, και εμείς ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, πάρα πολύ επικοδομητικά αυτά που μας είπατε και τώρα περνάμε σε ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Έχετε ε, κάτι να ρωτήσετε τον κύριο Ντικάρλο. Παρακαλώ. Τσίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Ντικάρλο, τον δόκτωρο Ντικάρλο για όλα αυτά που μας είπε και από ό,τι ακούσαμε, εσεί έχετε συγκεντρώσει πολύ σημαντική και πολύτιμη εμπειρία. Ε, τώρα, όσον αφορά τα βασικά θέματα της ε, δουλειάς του γραφείου, της ιδιοκτησίας, της ε, ε, διανοητικής ιδιοκτησίας. Εσείς έχετε στόχο να στηρίξετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, κυρίως μέσω της κατεγραφής, κάτι που κατά την άποψή μου εκεί παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Αναφερθήκατε στον αθέμητο ανταγωνισμό. Πρέπει να έχουμε κατανοού ότι όταν πρόκειται για παραποιημένα προϊόντα, δεν είναι μόνο το νομικό θέμα, οι δυσκολίες που προκύπτουν σε σχέση με την απασχόληση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές φορές θέματα που έχουν σχέση και με την υγεία των εργαζομένων. Έχουμε κατά νου τα παιχνίδια, τα καλλιντικά και πάρα πολλά άλλα. Άρα δηλαδή είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Και θίξατε και άλλο ένα θέμα, το θέμα του συντονισμού με τις εθνικές αρχές για να αποφεύγεται η παραποίηση και ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις που δουλεύουν πάνω σε αυτό το θέμα, όπως επίσης και στο θέμα της τεχνολογικής καινοτομία. Αυτά που μας είπατε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, έχοντας κατά την εμπειρία εμπειρία σας, ε, γιατί μιλάμε για απειλές όχι μόνο οικονομικές, αλλά και απειλές που αφορούν την υγεία των εργαζομένων. Εσείς ε, πώς πιστεύετε ότι μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικά τα μέτρα, αλλά και οι πρωτοβουλίες για τις οποίες μας μιλήσετε. Δηλαδή, αν θέλετε, πώς ε, μπορούμε να βελτιώσουμε καλύτερα τις δικές μας παρεμβάσεις και να βελτιώσουμε καλύτερα και τις παρεμβάσεις του το γραφείο της διανοητικής ιδιοκτησίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως ε, μπορώ και εγώ να μιλήσω Ιταλικά. Χαίρομαι πάρα πολύ Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, ε, πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι η συνεισφορά του δικού μας του γραφείου μπορεί να λάβει χώρα σε τρία επίπεδα. Πρώτον, ευαισθητοποίηση σε πολιτικό επίπεδο, γιατί πιστεύω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Από δικής μας ε, πλευράς ε, ξεκινήσαμε μέσα από το παρατηρητήριο για τα θέματα τα δικά μας. Συνεργαζόμαστε με τον ΟΑΣΑ για να καταρτήσουμε μελέτες που θα αποδεικνύουν ποιες είναι οι επιπτώσεις της παραποίησης τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι αλήθεια ότι όταν μιλάμε για την παραποίηση ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί το αντιμετωπίζουν ως ένα πλημέλημα, ότι είναι κάτι που δεν είναι και τόσο σημαντικό, ενώ έχει πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση και σε άλλα θέματα, παρεμφερεί. Εγώ πιστεύω, όπως είπατε και εσείς, ε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικής φύσεως. Ε, πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε, να εξηγήσουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις στην απασχόληση, αλλά υπάρχουν, όπως είπατε, και κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ακόμα ότι η παραποίηση αφορά μόνο τη μόδα και τα προϊόντα της μόδας. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα προϊόντων παραποιημένων που ε, φέρνουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Εμείς ως γραφεία, γραφείο αρχίσαμε να κάνουμε κάποιες αναλύσεις και στο επόμενο στρατηγικό σχέδιο θέλουμε να εμβαθύνουμε σε αυτά τα θέματα. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι επίσης σημαντικό και πρόκειται για μια στρατηγική συνεργασία που ε, θέλουμε να θεσπίσουμε με τη Europol. Είναι το θέμα των ε, ε, εγκληματικών ομάδων που συνδέονται με την παραποίηση και θεωρούν ότι η παραποίηση είναι κάτι πολύ ελκυστικό, ότι από πλευράς ποινική δεν συνεπάγεται και δεν έχει τους ίδιους κινδύνους, όπως παραδείγματο χάρη το εμπόριο των ναρκωτικών. Ε, με την Europol θέλουμε να συνεργαστούμε, να συγκεντρώσουμε πληροφορίες και να αναδείξουμε σε πολιτικό επίπεδο ε, τους ε, υπεύθυνου και να αναδείξουμε και τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην παραποίηση και τις εγκληματικές ομάδες. Τώρα, κάτι άλλο. Το θέμα είναι να ενταθεί ο έλεγχος. Έχουμε τα τελωνία, την αστυνομία που κάνουν βέβαια πάρα πολύ καλή δουλειά. Η παραποίηση ε, δεν ε, ήταν προτεραιότητα και δεν υπάρχουν πάρα πολλά κονδύλια για να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της. Άρα δηλαδή ε, πρέπει να κάνουμε καλύτερη χρήση των κονδυλίων που υπάρχουν, να καταλήγουμε σε καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων. Ε, επειδή σας μίλησα για τη συνεργασία με τη Europol, εμείς θέλουμε να υπάρχει ένα ε, σύστημα ε, το οποίο θα επιτρέπει τη συνεργασία με τη Europol για την αντιμετώπιση της παραποίησης. Θέλουμε στο επόμενο στρατηγικό σχέδιο να υπάρχει ένα είδος hub, ένας κόμβος για να αντιμετωπίζεται η παραποίηση και με τον τρόπο αυτό να στηρίζονται οι διάφορες εθνικές αρχές. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η τεχνολογία. Αναφερθήκατε και εσείς σε αυτήν. Ε, να χρησιμοποιήσουμε την ε, τεχνολογία. Ε, μίλησα για αυτή την πρωτοβουλία, το Φόρουμ Αντιμετώπισης της Παραποίησης. Ξέρετε, πολύ σημαντικό είναι η ενημέρωση γιατί πρόκειται για καθαρά τεχνικά θέματα, άρα δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν και απαραίτητες δυνατότητες αντιμετώπισης. Και η δικαιοσύνη και εκείνη ε, πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Με τη EuroJet ε, έχουμε φτιάξει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ε, υπουργείων που ασχολούνται με το θέμα και προτιθέμεθα να οργανώσουμε και ένα workshop για τους δικαστές για να ενημερωθούν και αυτοί. Σημαντικά όλα αυτά, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το θέμα της ζήτησης για τα παραποιημένα προϊόντα. Σε τελική ανάλυση, αν υπάρχει αυτό το φαινόμενο, είναι διότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να αγοράζουν ε, παραποιημένα προϊόντα και γι' αυτό θα πρέπει να οργανώσουμε εξτρετίες που θα επιτρέπουν ε, στους ε, καταναλωτές να κατανοήσουν ότι η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας για τη τελική ανάλυση όλα αυτά σημαίνουν ε, καινοτομία και μέλλον για τις επιχειρήσεις, άρα και μέλλον για τους νέους μας και για τους εργαζόμενους. Αυτά θα σταματήσω εδώ, αλλά όπως βλέπετε το θέμα αυτό είναι ένα θέμα που με παθιάζει, ίσως και γι' αυτό να μακρηγόρησα και λιγάκι. Έχουμε άλλους ε, τρεις ομιλητές ε, που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις ε, και θα δεχτούμε τώρα όλες τις ερωτήσεις γιατί τελείως δεν θα έχουμε πια χρόνο. Παρακαλώ και στις επόμενες απαντήσεις ή δυνατόν να είσαστε πιο σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στανκανέλη. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Διάβασα το βιογραφικό σας και διάβασα και το διαγραφικό της κυρίας Χέρμαν. Άκουσα αυτά που μας είπατε, πολύ ωραία. Θέλω όμως να κάνω μία ερώτηση. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε γιατί πιστεύετε ότι μπορείτε να αναπτύξετε καλύτερα το ρόλο που επιθυμείτε από την συνυποψήφιά σας. Κυρία Μέλχερ, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και για τις ε, πληρέστατες απαντήσεις σας. Είπατε ότι είναι σημαντικός ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πώς βλέπετε ότι θα είναι δυνατόν να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησία δεν θα χρησιμοποιηθούν για να μπλοκάρουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν θα έχουν καταχωρήσει ε, δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας. Πώς θα τις προστατεύσουμε από μεγάλες ε, επιχειρήσεις ε, που είναι εδρεωμένε στην αγορά. Η καταχώρηση ενο σήματος ή ενό υποδείγματο είναι μια δαπανηρή διαδικασία. Πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, να αποκομίσουν τα ωφέλη από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ε, αναφέρεται με υπερηφάνεια ότι αυτοχρηματοδοτείται το γραφείο και είναι και ο μεγαλύτερος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ανησυχεί λίγο ε, μήπως επιβαρύνουμε τις εταιρείε μας κατά αυτόν τον τρόπο που τις υποχρεώνουν υποχρεώνουν τα πνευματικά τους δικαιώματα δεν το θεωρώ αυτό σκοπό το να έχουμε ένα τεράστιο γραφείο διανοητική ιδιοκτησία στο Αλικάντε. Πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτού του θέματος. Ακόμη είχα τη χαρά να συμμετάσχω στη συζήτηση για, το, για τα ευρωπαϊκά δικαιώματα ιδιοκτησίας. Κάναμε μια τέτοια ε, συζήτηση στη Δανία και το επιχείρημα υπέρ είναι ότι ε, πολλές φορές στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά δικαιώματα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Πώς μπορούμε να έχουμε ε, καινοτομία και να μην πνίγεται η καινοτομία μέσω των απαιτήσεων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων διανοητικής διοκτησίας πώς μπορεί να εξασφαλίζεται. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το προσωπικό του γραφείου του οργανισμού, του γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας, πώς θα φροντίσετε να εξασφαλίζετε το προσωπικό έναντι περιστατικών παρενόχλησης. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ξεπεράσατε το χρόνο σας, οπότε δίνω το λόγο ε, και στον επόμενο μιλητή για μια ερώτηση ακόμη πριν απαντήσει ο κύριος Ντικάρλο. Ευχαριστώ πολύ. Πολλέ από τι προκλήσει για τι παραβιάσει διανοητική διοκτησία προέρχονται από τρίτε χώρε και συγκεκριμένα πολλέ από την Κίνα. Έχετε σχετική εμπειρία για συνεργασία με την Κίνα και πώ νομίζετε μπορεί να συνεισφέρει το γραφείο σε αυτό το τομέα. Δεύτερο ερώτημα. Κατά τη γνώμη σας, Μπορεί το γραφείο να κάνει κάτι συγκεκριμένο για να βοηθήσει τους κατόχους δικαιωμάτων δικαιω... διανοητικής ιδιοκτησίας ε, έναντι της ε, κυβερνοπειρατείας και άλλων προκλήσεων από το διαδίκτυο. Αν μπορείτε να είστε σύντομος, μέσα σε τρία λεπτά να με δώσετε τις απαντήσεις σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας γιατί που με ρωτήσατε γιατί πιστεύω ότι μπορώ να κάνω καλή δουλειά ως αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής. Νομίζω το εξήγησα και στο τέλος της ε, παρέμβασής μου. Σας είπα ότι έχω συγκεντρώσει ευρύτατη εμπειρία από πολύ σημαντικές δραστηριότητες του γραφείου μας. Άρα δηλαδή έχω έτσι ένα φάσμα ε, που μου επιτρέπει να γνωρίζω τι γίνεται στο γραφείο, στο εσωτερικό, ε, έξω από αυτό. Έχω και τη δυνατότητα να κατανοήσω ποιες είναι οι προκλήσεις του σήμερα αλλά και του αύριο και να μπορέσω να ε, δραστηριοποιηθώ για να αντιμετωπίσω τις ε, προκλήσεις. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι, κάτι, ε, είναι το εξής. Προσπάθησα να δραστηριοποιηθώ σε διεθνές και πολυπολιτισμικό επίπεδο και πλαίσιο. Αυτό είναι αυτό που χαρακτηρίζει το γραφείο μας. Μέχρι τώρα Υπάρχουν διάφορες ε, φάσεις που έχουν ε, ξεκινήσει. Ε, όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία, εξελέγην ως η καλύτερη επιλογή. Μετά ακολούθησαν διάφορες συνεντεύξεις. Ήταν όλοι υπέρ της υποψηφιότητάς μας και αυτό αποδεικνύει ότι έχω καλή εμπειρία και αυτό πιστεύει και ο εκτελεστικός διευθυντής. Τώρα, όσον αφορά το δικό σας ερώτημα, ε, θέλω να πιστεύω ότι ε, απάντησα σε όλα, αλλιώς πέστε μου αν ξέχασα ή αν θα ξεχάσω τώρα κάτι. Όσον αφορά το γεγονός ότι η καταγραφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να είναι δαπανηρή, θα ήθελα να σας πω επ' αυτού ότι το γραφείο μας ε, δύο φορές ε, μείωσε τις εισφορές που καταβάλουν επιχειρήσεις για να καταγράψουν, να καταχωρήσουν μάλλον ε, τα δικαιώματα copyright. Ε, το επέτρεψε αυτό βέβαια ο προϋπολογισμός μας, αλλά και κυρίως εμείς θέλαμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις ε, να καταχωρήσουν τα δικαιώματά τους, το copyright. Ε, το να υπάρχει κακή χρήση ε, της διανοητικής ιδιοκτησίας. Ε, αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα bullying, ένας εκφοβισμός ε, που λαμβάνει η χώρα σε σχέση με τη διανοητική ιδιοκτησία. Πράγματι λοιπόν εξετάζουμε όχι μόνο το πώς μπορούμε να υπερασπιστούμε καλύτερα την διανοητική ιδιοκτησία, αλλά και πώς μπορούμε να αποφύγουμε, να παρεμποδίσουμε το bullying, τον εκφοβισμό που είναι πρόβλημα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λαμβάνουν επιστολές από μεγάλες εταιρείε και το εξετάζουμε αυτό. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά θέματα που έχουν τεθεί. Φοβάμαι ότι πρέπει να σταματήσετε. 30 δευτερόλεπτα, τα τελευταία δευτερόλεπτα ε, για την τελευταία απάντηση. Λοιπόν, έχω εμπειρία σε θέματα διεθνούς ε, συνεργασίας. Ήμουνα αρμόδιος ε, για θέματα συνεργασίας με την Κίνα και σε αυτό το πλαίσιο συνεργάστηκα με διάφορους τρόπους η συνεισφορά του γραφείου όπως είπα και προηγουμένως το να βοηθήσει όσους χαράσουν πολιτική ε, να ε, συγκεντρώσουν πληροφορίες και δεδομένα και επίσης ε, και να διασφαλίσουν ότι θα υπάρξει βελτίωση προ όφελο ε, των ε, μικρομεσαίων επιχείρησεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δραστηριοποιούνται στην Κίνα. Και αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει και συνεργασία στην Ευρώπη έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα παραποιημένα προϊόντα που έρχονται από την Κίνα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για να επεκταθώ περιττέρω. Ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας και ζητώ συγγνώμη που χρειάστηκε να σας σταματήσω, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε με τη διαδικασία. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Χάρμαν για μια παρουσίαση 10 λεπτών και θα έχετε και στη συνέχεια χρόνο για τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Thank you, Madam Chair, honorable members of the Parliament. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι ο σκοπός του γραφείου, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Θέτω την ερώτηση και την απαντώ μόνη μου. Ο σκοπός είναι να υπηρετεί το κοινό ως κέντρο αριστείας για τη διανοητική ιδιοκτησία, για να βοηθά τις επιχειρήσεις. Ας δούμε λοιπόν πώς τα πάει το γραφείο. Όπως ακούσαμε, πάει πάρα πολύ καλά. Αυξάνονται οι αιτήσει, ο αριθμό αυξάνεται κάθε χρόνο. Αυξάνονται και τα συνολικά έσοδα, αλλά και χάνει χρήματα. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, κάθε χρόνο έχει ζημίες 1,5 εκατομμύρια γιατί τα χρήματα παραμένουν ανενεργά σε τράπεζες έχουν παραταθεί οι χρόνοι καταχώρησης, αν το συγκρίνουμε με το 2017. Η ικανοποίηση των πολιτών έχει μειωθεί, αρκετά θα έλεγα, από 92% σε 85% και το ποσοστό επιβεβαίωση των αποφάσεων στο Γενικό Δικαστήριο έχει μειωθεί από 86% σε 77%. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο Ας δούμε και ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο σε ολόκληρο τον κόσμο γύρω από το γραφείο. Υπάρχουν νέοι τρόποι εργασίας, οικονομία του διαμερισμού, διαμοιρασμού, συγγνώμη, κυκλική οικονομία. Υπάρχουν επίσης νέοι τρόποι κατανάλωσης, συμβόλαια τα οποία συνάπτονται διαφορετικά, συνειδητοί καταναλωτές, ιδίως οι νέοι. Συνειδητοί καταναλωτές όπως εγώ που δεν χρησιμοποιούμε πλαστικό και έχουμε το θερμός μας μαζί μας. Έχουμε δει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι περιμένουν ένα διαφορετικό ρόλο από τα γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας, όχι μόνο την καταχώρηση δικαιωμάτων, αλλά και υποστήριξη και καθοδήγηση. Και βέβαια υπάρχει και η τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, πολύ διαφορετικοί τρόποι χρήσης της τεχνολογίας και είναι πολύ γρήγορη η εξέλιξη. Τώρα, ας δούμε το γραφείο πιο προσεκτικά. Ποιες είναι οι προκλήσεις. Βεβαίως, η συνεχιζόμενη εφαρμογή της μεταρρύθμισης για τα σήματα. Αυτό απασχολεί ιδιαίτερα το γραφείο και κάποια από τα ανησυχητικά στοιχεία προκύπτουν λόγω της μεταρρύθμισης των σημάτων. Υπάρχουν και νέα καθήκοντα, ιδίως η αναθεώρηση του κανονισμού για τα σχέδια και υποδείγματα και μια πιθανή πρωτοβουλία για τις μη, γεωγραφι... μη γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις. Η τεχνητή νοημοσύνη και πάλι και εδώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει ευθύνη σε αυτόν τον τομέα. Δραστηριότητες επίσης σε διεθνές επίπεδο μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας αλλά και σε άλλους οργανισμούς. Και όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι διασυνοριακές γιατί είναι ε, κάτι το οποίο δεν έχει σύνορα η διανοητική ιδιοκτησία. Ε, ε, δυστυχώς υπάρχουν και οι παρατυπίες και οι περιπτώσεις απάτης, οι οποίες επίσης δεν έχουν σύνορα. Και η συνεργασία λοιπόν μεταξύ των δικαστικών αρχών και των διοκτικών αρχών και άλλων οργανισμών παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Το στρατηγικό σχέδιο τώρα. Ακούσαμε ήδη για το στρατηγικό σχέδιο. Εδώ νομίζω ότι υπάρχουν τρεις βασικοί στόχοι. Καταρχήν, αξιόπιστο σύστημα διανοητικής ιδιοκτησίας και κατά μένα αυτό σημαίνει συνεργασία. Συνεργασία μεταξύ των εμπειρογνωμόνων από διαφόρους οργανισμούς που θα πρέπει να ανταλλάσσουν εμπειρίες και γνώσεις, συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, εθνικών γραφείων και ευρωπαϊκού γραφείου, για την ενίσχυση του επίπεδου εξυπηρέτησης και συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους, γιατί πρέπει να ακούμε τις ανάγκες τους, να ακούμε τι χρειάζονται. Υπηρεσίες επικεντρωμένες στον πελάτη. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό καθήκον. Σήμερα αυτό σημαίνει κυρίως ε, χρήση τεχνολογίας για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ε, και δεν πρόκειται μόνο για την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πολλές άλλες λύσεις. Μιλήσαμε για την τεχνολογία λυσίδα στοιχειών, το blockchain. Θέλουμε να υπάρχει τεχνολογία περισσότερο κατανοητή και ευέλικτη και φτιαγμένη στα μέτρα του καθενός. Χρειάζεται καλύτερη διοίκηση. Χρειαζόμαστε ε, ανθρώπους με ενθουσιασμό για να έχουμε ένα ισχυρό οργανισμό με ανθρώπους που θα έχουν ε, ταλέντο, που θα τους κρατήσουμε, που θα τους αναπτύξουμε στο πλαίσιο ενός ε, διαφανούς οργανισμού. Τώρα, πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω σε όλα αυτά. Υπηρέτησα το κοινό στην Εστονία επί 25 χρόνια. Στην Εστονία υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης και χρήσης ε, πολλών ε, τεχνολογικών ηλεκτρονικών λύσεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20 ε, τέτοιες λύσεις, συστήματα που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, που λειτουργούν στο δημόσιο τομέα στην Εστονία, που καθημερινά εξυπηρετούν τους πολίτες. Προσωπικά έχω εμπειρία με τη δημιουργία τέτοιων συστημάτων ηλεκτρονικών και ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται για τον επανασχεδιασμό του τρόπου εργασίας, είναι για την επανεκκίνηση του τρόπου σκέψης. Θέλουμε να είμαστε ενεργοί, να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για τις υπηρεσίες, τις οποίες αποκαλούμε αόρατες υπηρεσίες. Δηλαδή πρέπει συνεχώς να γνωρίζουμε τις επιθυμίες των πολιτών, των καταναλωτών, χωρίς να έχουμε στερεότυπα. Και αυτό προκύπτει από την εμπειρία. Πρέπει να ξέρουμε τι είδους δεδομένα δίνουμε στο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για να το κάνουμε να λειτουργήσει και για να μπορέσει να μάθει. Ένα αξιόπιστο σύστημα διανοητικής ιδιοκτησίας. Συνδυάζω πήρα και ε, στα θέματα διοίκησης και ως δικαστής. Επί 20 χρόνια και παραπάνω ε, είμαι στο νομικό τομέα και έχω εμπειρία σε θέματα και δημόσιου τομέα και ε, δικαστικού σώματος. Ασχολούμαι με την τεχνητή νοημοσύνη και με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Εσθονίας. Οι δεξιότητές μου καλύπτουν ευρύ φάσμα ε, στην εκπαίδευση φοιτητών και σε πανεπιστήμια και σε άλλες μορφές εκπαίδευσης και έχω πολλές δεξιότητες για την επίλυση διαφορών και νομικών διαφορών όπως και για την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και στην Εσθονία και σε διεθνές επίπεδο. Έχω ζήσει όλη μου τη ζωή σε κοινωνίες που αλλάζουν. Σας υπενθυμίζω ότι γεννήθηκα στη Σοβιετική Ένωση. Άρα οι αλλαγές και η καινοτομία για μένα δεν είναι κάτι καινούριο, δεν φοβάμαι την αλλαγή. Αναδιάρθρωσα το ε, Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της Εσθονίας. Έχω εργαστεί σε πολλές στρατηγικές επιτροπές για την ε, μεταρρύθμιση της Εστονίας, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για νέους τρόπους εργασίας και για στρατηγικό προγραμματισμό για την τεχνητή νοημοσύνη. Και έχω πραγματικά προσωπική εμπειρία στην Εστονία. Έχουμε πολλά ε, πιλωτικά προγράμματα. Είμαστε τόσο φτωχή χώρα που δεν μπορούμε κατευθείαν να μπούμε σε μια μεγάλη πρωτοβουλία και να δαπανίσουμε πολλά δημόσια κονδύλια για κάτι το οποίο δεν είμαστε σίγουροι ότι δουλεύει. Οπότε έχουμε πολλά πιλωτικά προγράμματα. Ξεκινάμε, δοκιμάζουμε, βελτιώνουμε και μετά το εφαρμόζουμε σε δημόσιο, στο δημόσιο τομέα με συγκεκριμένες λύσεις. Πρέπει να ολοκληρώσω, μου λέει η Πρόεδρος. Φτάνω στο τέλος της ομιλίας μου τονίζω ότι είμαι υπέρ της διαφάνειας ε, και ε, είμαι υπέρ του σκανδιναβικού τρόπου δουλειάς που σημαίνει υπευθυνότητα, λήψη αποφάσεων από τη βάση, ομαδική εργασία ώστε να εξασφαλίζω ισορροπημένη ηγεσία, ομαδικό πνεύμα δουλειάς, διαφορετική προσέγγιση και νέες ιδέες. Αυτά μπορώ να δώσω. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Ερωτήσεις τώρα. Η κυρία Μαρκιού πρώτα απ' όλα και μετά θα δούμε για τις επόμενες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Πραγματικά με χαρά βλέπω δύο υποψηφίους τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους να μας παρουσιάζουν την υποψηφιότητά τους. Εσείς μας μιλήσατε για το τι κάνετε στην Εστονία. Είδα στο βιογραφικό σας ότι έχετε εμπειρία και ότι έχετε εργαστεί ε, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα για τη συνεργασία σας ε, με το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και πώς θα υλοποιήσετε ε, το... και πώς θα μεταφέρετε το ρόλο που έχετε αναλάβει μέχρι τώρα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής ε, Ιδιοκτησίας και πώς η εμπειρία σας ε, στην Εστονία ε, μπορεί να σας εμπνεύσει και να σας βοηθήσει, να σας καθοδηγήσει στα νέα σας καθήκοντα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας ώστε να λειτουργήσει και αυτό τόσο καλά όπως η εστονική δίκηση και πώς θα συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ιδιωτική Διοκτησία. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Η... Μιλάτε για την εμπειρία μου στο Εστονικό Γραφείο Διπλωμάτων ευρεσιτεχνία ή στο Ευρωπαϊκό. Ήμουν μέλος του Συμβουλίου Προσφυγών που είναι κάτι σαν εθετίο, Αν παραλύσουμε το σύστημα με το δικαστικό. Αυτό σημαίνει ότι συζητούνται εκεί πολύ σημαντικά νομικά ζητήματα. Συμμετείχα, λοιπόν, νομίζω, σε δύο ή τρεις διαφορετικές υποθέσεις που είχαν να κάνουν με ε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Κάτι το οποίο βρήκα πάρα πολύ σημαντικό γιατί η βιοτεχνολογία είναι κάτι που έχει να κάνει με το μέλλον, είναι η επιστήμη του μέλλοντος ήδη από τώρα. Η εμπειρία μου στην Εστονία, ρωτάτε, κοιτάξτε κάθε εμπειρία ε, μπορεί να είναι χρήσιμη. Και το δικό μου δυνατό σημείο γενικά είναι ότι ξέρω να ακούω τους ανθρώπους. Ακούω και είμαι σε θέση να καταλάβω τις ανάγκες τους. Από την άλλη είμαι ιδιαίτερα επίμονη να έχω αποτελέσματα. Στην Εστονία μου πήρε τέσσερα χρόνια για να καταφέρω να κάνω τους πολιτικούς να κατανοήσουν την ανάγκη για να αναδιοργάνωση. Αναδιάρθρωση ενός γραφείου είναι κάτι το οποίο είναι πάντα επίπονο. Ακόμα κι αν είναι για το καλό, είναι δύσκολο. Χρειάζεται λοιπόν κατανόηση για την άλλη άποψη και δυνατότητα να εξηγήσει κανείς το τι χρειάζεται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορώ να κάνω. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Α, η Κάραν πάλι. Ίσως ήμουνα αδική και δεν σας ρώτησα ε, τα ίδια πράγματα όσον αφορά ε, το οικονομικό βάρος που πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν πρόκειται για τη δικιά τους πνευματική ιδιοκτησία. Υπάρχουν νομικά μέτρα, όπως υποχρεωτικές άδειες, Οπότε πιστεύω ότι το ένα πράγμα είναι ότι η νομοθεσία πρέπει να διαθέτει ισορροπημένα μέτρα προκειμένου να ενισχύει την καινοτομία. Να μην τη σταματάει, να μην την εμποδίζει. Από την άλλη μεριά πιστεύω ότι είναι εξίσου σημαντικό ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δίνουμε τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις δικές του λύσει διανοητική ιδιοκτησία. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσω χρηματοδότηση ή μπορεί να γίνει μέσω ευκαιριών που τους δίνουμε να συμμετέχουν σε hackathons ή σε άλλες τέτοιες δομές. Είναι όμως και θέμα συνειδητοποίησης. Εγώ πραγματικά πιστεύω στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Και υπάρχουν ε, πραγματικά πολλές δυνατότητες, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να χρησιμοποιήσουν λύσεις οι οποίες εύκολα έχουν άδεια, χωρίς να κοστίζουν ακριβά από την άλλη, ναι, μιλάμε για χρήματα, έτσι. Στον κανονισμό που διέπει τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας υπάρχει διάταξη που λέει ότι κάποια από τα χρήματα αυτά τα οποία συλλέγονται από τις επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέφουν στις χώρες μέλη. Και δεν νομίζω ότι σπαταλά χρήματα το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής ε, Ιδιοκτησίας. Όχι, τα χρησιμοποιεί για τις επιχειρήσεις. Μιλάμε για τις δραστηριότητες του παρατηρητηρίου εδώ. Και επίσης για τη δημιουργία δικτύων χρηστών ή εμπειρογνωμόνων στην ε, εκπαίδευση και την κατάρτιση, πράγματα από τα οποία εποφελούνται οι επιχειρήσεις έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε πολύ λέει Πρόεδρος. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, οπότε ήθελα να ρωτήσω... Α, εσείς, παρακαλώ, η κυρία Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ζητώ συγγνώμη ε, γιατί θα είμαι η τελευταία και επιμένω, αλλά θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Χερμάν ε, για την ε, παρουσία της και να τη συγχαρώ για την εμπειρία. Στα γρήγορα όμως μια ερώτηση, περίπου τα ίδια όπως αυτά πρότισα και τον προηγούμενο υποψήφιο. Η διανοητική ιδιοκτησία ε, και σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη που θίξατε εσείς ε, ε, και που συνεπάγεται πάρα πολλές δυσκολίες και προκλήσεις έχει σχέση και με την παραποίηση των προϊόντων. Το αναφέρετε και εσείς, το επενυχτήκατε. Θέλω να ρωτήσω πώς μπορεί το γραφείο να παρέμβει έτσι ώστε να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο και σε διεθνές επίπεδο. Γιατί ελέγχθηκε προηγουμένως ότι ε, αυτό το φαινόμενο δεν υπάρχει μόνο στην Ευρώπη αλλά γενικότερα σε διεθνές επίπεδο. Θέλω λοιπόν να μας πείτε πώς πιστεύετε ότι μπορείτε, μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δώσατε τη δυνατότητα να κάνω αυτή την ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας συμμετέχει σε διάφορα δίκτυα, διεθνή δίκτυα, τα οποία ασχολούνται με θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και θέμα, με θέματα παραποίησης προϊόντων. Όπως είπα και πριν, εγώ πραγματικά πιστεύω στην εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι η συμμόρφωση στο νόμο είναι κάτι το οποίο μπορεί να μάθει κανείς με την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση. Οι χρήστες δηλαδή θα έπρεπε να διαπαιδαγωγηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και οι διεθνείς συνθήκες που υπάρχουν λειτουργούν μέσα από θεσμούς και από ανθρώπους. Και αυτό είναι ο κρίκος που συνδέει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας με ε, την ε, ζωή που μπορούν να αποκτήσουν αυτές οι διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ε, δεν υπάρχει άλλο χέρι που να βλέπω. Εντάξει, τότε ας περάσω στη δικιά μου την ερώτηση που έχει να κάνει και με αυτό που είπατε τώρα πόσο πιστεύετε ακριβώς την εκπαίδευση, στην ε, κατάρτιση ότι μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή. Μπορείτε να εξηγήσετε το ρόλο του copyright, πώς το εξηγεί κανείς και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας φροντίζει να μάθει στον κόσμο ποια είναι η σημασία του copyright. Το κάνει ή θα το κάνει στο μέλλον, θα φροντίσετε να το κάνει. Απάντηση. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διονυτικής Ιδιοκτησίας θα ασχοληθεί και με νέα καθήκοντα και αρμοδιότητες πολύ σύντομα. Υπάρχει το πακέτο για το copyright που δημοσιεύθηκε την Άνοιξη. Και πιστεύω ότι αν θέλουμε το Ευρωπαϊκό Γραφείο διονοτική Ιδιοκτησίας να καταστεί ένας κόμβος αριστείας, θα πρέπει πράγματι να ασχοληθεί και με το copyright. Ε, βέβαια δεν υπάρχει καταχώρηση και είναι πολύ πιο περίπλοκο το θέμα. Αλλά έτσι κι αλλιώς πρόκειται για ένα βήμα προκειμένου να καταστεί το γραφείο Κόμβος Αριστείας. Ε, πιστεύω πως ναι, είναι δυνατόν και είναι μάλιστα αναγκαίο να συνδέσουμε το copyright με το χαρτοφυλάκιο αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε. Κυρίως αν μπορώ να το συγκρίνω με την εμπειρία μου όταν ήμουν δικαστής, που ήμουν δικαστής για την διανοητική ιδιοκτησία, ασχολούμασταν με το copyright, με τα σχέδια. Πάντα υπάρχει ή μπορεί να υπάρχει θέμα copyright όταν εξετάζει κανείς τέτοια ζητήματα σχεδίων και αν υπάρχει δίωξη με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πάντα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Το ποιος είναι ο ιδιοκτήτη. Ποιο κατέχει αυτήν την διανοητική ιδιοκτησία. Οπότε ναι, ναι, σίγουρα θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό, εφόσον αναλάβω τα καθήκοντά μου. Πρόεδρος, ωραία, δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο που ήρθατε εδώ και απαντήσατε στις ερωτήσεις μας. Τίποτα άλλο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Για δύο λεπτά θα κλείσουμε γιατί μετά θα ξαναρχίσουμε τη συνεδρίασή μας και